Colleagues, if I could uh, start Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλημέρα. Ξεκινάμε τις πρωινές μας εργασίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Σιδηροδρόμων, τον κύριο Βεσλάιτ, που είχε την καλοσύνη να έρθει και την έμψα μετά. Τον κύριο Ντιρόιτε σίγουρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα το αγώνα, ζητώντας από τον εκτελεστικό διευθυντή του ERA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδοδρόμων, να μας μιλήσει και μετά ελπίζω να καταφτάσουν και άλλοι συνάδελφοι, να τα καταφέρουν να περάσουν το χιόνι και μπαίνω στον πειρασμό να λέω αστιάκια για τα διάφορα είδη λάθος είδος χιονιού αλλά οι σιδηροδρομικοί στενοχωριούνται μας μιλήσουμε για το λάθος είδος χιονιού. Έχετε... Λοιπόν θα καταστεί. Κύριε Βέσλα, πήγα να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο και μου άφησαν αυτό το σημειωματάκι. Μάλλον για το web streaming χρησιμοποιείτε αυτό το μικρόφωνο και μου έστειλε αυτό το διακριτικό σημειωματάκι που βλέπετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βέσλα. Έχουμε μια περιορισμένη παρουσίαση κάποιες ε, διαφάνειες ε, που θα δείξουμε με το PowerPoint. Έχω, έχω την ευχαρίστηση να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την εξέλιξη των, ε, της υπηρεσίας μας, της υπηρεσίας σιδηροδρόμων. Είμαστε στον έκτο. Θα μπούμε. Μπήκαμε στον έκτο χρόνο ύπαρξης της υπηρεσίας και έχουμε κάνει πολλέ δραστηριότητε. Η διαφάνεια που ήθελα να παρουσιάσω σαν πρώτη ήθελα να σα δείξει ότι ένα από τα ωφέλη τη υπηρεσία, ακόμα και δεν είναι εύκολο να το χειριστούμε, είναι ότι η μόνη στην Ευρώπη όπου συναντώνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και ήθελα να σας δείξω με τι πράγμα δουλεύουμε τι γίνεται τυποποίηση, έρευνα, βιομηχανία, επιχειρήσει του σιδηροδρόμων, υποδομέ των σιδηροδρόμων, διαχειριστέ των υποδημών σιδηροδρόμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, εθνικέ υπηρεσίε ασφαλεία, η υπηρεσία TNT, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει τομέα τη ευρωπαϊκή οικονομία που έχει τόσου φορεί όσο οι σιδηρόδρομοι. Του καλωσορίζουμε όλου. Στην ε, υπηρεσία έχουμε 12 σημαντικές δραστηριότητε που ασκούμε. Πρώτη προτεραιότητα είναι το θέμα της ασφάλειας. Πρέπει να αναπτύξουμε τα συστήματα διαχειρίσεως της ασφάλειας, τις μεθόδους, τις αρχές, τον έλεγχο, διερεύνηση ατυχημάτων. Είχαμε δυστυχώς κάποιες δυνατότητες να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Ε, κανονισμοί, ρύθμιση και επιστοποίηση είναι σημαντικό όχι μόνο εναρμόνιση αλλά και ανάπτυξη κοινών συστημάτων ε, ε, πιστοποίησης, ο έλεγχος των επιδόσεων ασφαλείας, υποβολή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμογή της οδηγίας, όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από μοτίμους έλεγχος και ανάπτυξη έλεγχου, διασταυρούμενο έλεγχο μεταξύ των εθνικών αρχών ασφαλείας διαλειτουργικότητα. Έχουμε ετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργικότητα και έχουμε πάρα πολλή δουλειά συντονισμού με του φορεί τυποποιήσεω, SENSE, ENELEC και έτσι. Και επίσης έχουμε και προτάσεις για τους μηχανοδηγού των τρένων, πιστοποίηση, κατάρτιση, κέντρα κατάρτισης και τι καθήκοντα θα έχει το υπόλοιπο προσωπικό των σιδηροδρόμων. Ελέγχουμε τη λειτουργικότητα. Δημοσιεύσαμε με μεγάλη επιτυχία κάτι που το λέπισα στη σελίδα, την πρώτη έκθεση δηλαδή, όσον αφορά τη διελειτουργικότητα. Προμηνών το δημοσιεύσαμε. Παρακολουθούμε την τεχνική αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων και του ε, φορεί κοινοποίησεω και έχουμε σημαντικό ρόλο για τι διάφορε αδειοδοτήσει και καθορίζουμε, βλέπουμε ποιοι είναι οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζουμε. Και έχουμε και την αρχή ETRMS, είμαστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ETRMS και τις μεθόδου αξιολογήσεως συμμόρφωσης. Έχουμε πολλά μητρώα βάσης δεδομένων, με άδειε χαρακτηριστικά των σιδηροδρόμων, των βαγονιών κλπ. Έχουμε μικρή μονάδα ω οικονομικής, οι οποίε αυξάνονται βέβαια. Ελέγχουμε μεθοδολογία και την εκ των προτέρων και των υστέρων ε, αξιολόγηση. Και επίσης έχουμε και πολλά άλλα καθήκοντα συμπληρωματικά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουμε 12 βασικές δραστηριότητε, αλλά μόνο 157 ε, καθήκοντα μας ανετέθησαν και έχουμε 140 μέλη στο προσωπικό, άρα μεγάλο φόρτο εργασίας όπως καταλαβαίνετε. Όσον αφορά την ασφάλεια, το 2010-2011 θα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλα τα καθήκοντα προβλέπει η Οδηγία Περισφάλειας, κοινέ μέθοδοι, στόχοι και δείχτες για την ασφάλεια. Το ίδιο για τη δελειτουργικότητα Ολοκληρώνουμε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Πολλή δουλειά γίνεται σύντομη περίοδο με περιορισμένα μέσα όσον αφορά την αμοιβαία αποδοχή και στο ERTMS e ε, η περίφημη τελευταία εκδοχή ετέθησε ισχύ, είναι σταθεροποιημένη, είναι εκδοχή ε, και είναι έτοιμη για επενδύσεις. Πολύ μικρή ομάδα όμως μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να ετοιμάσει όλα και για το 2012 έχει πολλή δουλειά την 3.0.0, τη βασική γραμμή του ETRMS και αυτό ήταν πρόκληση. Θα σας δείξω υπέροχη διαφάνεια. Α σας τα πω. Χθε είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στη συνέντευξη τύπου του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο κ. Γκρέιτον ήταν εκεί, παρουσιάσαμε τη μελέτη για την αξιολόγηση των επενδύσεων των συνδρομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά με κάποια σφάλματα ήταν η παρουσίαση τεχνική φύσεω και στο τέλο μα έδειξε το περίφημο παράδειγμα των διαφόρων ε, το πίσω μέρος των τρένων κλπ. Θα έπρεπε να σας δείξω τα 21 συστήματα που είχαμε. Από τον Ιούνιο έχουμε συμφωνήσει να έχουμε δύο συστήματα αντί 21 που είχαμε. Το σύστημα με τις λάμπες και το άλλο με την πλάκα την αντανακλαστική. Είναι συμβολικό θα έλεγα, δεν είναι συμβολικό όμως. Κάναμε λεπτομερή ανάλυση με το τομέα τι γίνεται με την εφαρμογή αυτού. Περίπου 250.000 εμπορικά τρένα σταματούν στα σύνορα για να αλλάξουν τις λάμπες τους κλπ. Και, και θα μειωθεί αυτός ο αριθμός στα 70.000. Θέλουμε να προσπαθήσουμε ένα κοινό σύστημα, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Σας ξέφυγε η Ιρλανδία, λέει ο πρόεδρο, και τη Φιλανδία. Ναι, ναι. Εκεί δεν ε, κάναμε κάτι. The uh, Δεύτερο παράδειγμα με συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι το κόστος πιστοποίησης των διαφόρων οχημάτων των συνδρομικών. Ρίξαμε μια ματιά στο κόστος αδειοδότησης των σιδηροδρομικών των, των σειρμών και το κόστος ε, ανακάτως μέλος. Και ξέρω τα επιχειρήματα της UNIFE, έχουν δίκιο. Η πρώτη αδειοδότηση ενός οχήματος από τα πλά μέχρι τα τρένα υψηλής ταχύτητος κοστίζει από 0,1 μέχρι 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε πρόθεσμα, να το αλλάξουμε αυτό. Ο μέσος όρος της μέσης αδειοδότησης τα κράτη-μέλη, αν περάσει τα σύνορα, είναι 1,6. Και για τα σύγχρονα βαγόνια 10 διαφορετικές αδειοδοτήσεις. 16 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος αν θέλει κανείς να περνάει από 10 κράτη-μέλη. Στο πρόγραμμα εργασίας που συμφωνήσαμε τον τομέα, δηλαδή και τους σιδηροδρόμους και τη γενικότερη ευρύτερη βιομηχανία στον τομέα, δεν θα αλλάξει. Η διασυνοριακή αποδοχή είναι ένα μπάλωμα που περιμένει την μακροπρόθεσμη εναρμόνιση. Με πρόθεσμα θέλουμε να μειώσουμε, να κρατήσουμε το κόστος της πρώτης αδειοδότησης, το κρατήσουμε χαμηλά, να μειώσουμε λοιπόν το κόστος και συμπληρωματικών αδειοδοτήσεων στο 50%. 800.000 ευρώ, με άλλα λόγια, ανά είδος σήμερα. Φαίνεται περιορισμένο, 400 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομεί ο τομέας, σε μια 15 ετία. Είναι ένα πρώτο βήμα. Έχουμε συλλέξει τους εθνικούς κανόνες και έχουμε χιλιάδες κανόνες που μαζέψαμε. Η ομάδα μας λοιπόν ταξινομεί τους ε, κανόνες, τους συγκρίνει, προσπαθεί να θέσει κάποια ισοδυναμία. Είναι σαν ένα παζλ με 10.000 κομμάτια, αλλά καλά πάει η δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, έλαβα δύο, τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες δραστηριότητε μας. Πρώτα απ' όλα διερεύνηση, ε, διελεύκανση ατυχημάτων. Η υπηρεσία δεν έχει άμεση εξουσία, αλλά είμαστε βασικά συντονιστικός φορέας και φορέας διαμεσολάβησης. Συντονίζουμε τις εθνικές ερευνητικές αρχές, στην περίπτωση του Βελγίου, γιατί υπήρχε ένα ερώτημα γι' αυτό, την ημέρα του ατυχήματο που συνέβη λάβαμε επίσημο αίτημα από το Βελγικό Υπουργείο και τον Βελγικό Φορέα Έρευνας να τους βοηθήσουμε στην έρευνα. Στείλαμε λοιπόν την ίδια μέρα μία ομάδα να τους βοηθήσει όταν είχε συμβεί το ατύχημα. Πήγαμε στον τόπο του ατυχήματος και μας ζήτησε και το μια επιτροπή του Βελικού Κοινοβουλίου να αξιολογήσουμε την κατάσταση στο Βέλγιο. Το δεχτήκαμε, διότι είναι γενική αποστολή που μας ανετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για όλα τα κράτη-μέλη και δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας ε, τον Οκτώβριο. Συναγάγαμε κάποια συμπεράσματα. Ο πολύ νέος ερευνητικός φορέας του Βελγίου δεν είχε τα μέσα, δεν ήταν έτοιμος να κάνει τη δουλειά, δεν είναι αρνητικό αυτό που λέμε. Περίπου 50% των κρατών μελών έχουν το πρόβλημα και τα βοηθάμε ε, να αναπτύξουν τις σχετικές δραστηριότητες. Και δυστυχώς αργά θα έχουν στη διάθεσή τους τελικά τα μέσα που χρειάζονται. Το ETRMS ε, χειριζόμαστε την 230D, την εκδοχή που είναι νόμιμη ε, και σταθερή θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση κάποιων προηγουμένων συστημάτων στην εκδοχή αυτή, 230D, αλλά χρειάζεται συντονισμός. Ας πούμε, σαν μέρος μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές του λογισμικού και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Η νέα η βάση η 3.0.0 ε, αναπτύσσεται με διαφανή τρόπο και πρέπει να είναι συμβατή με προηγούμενα συστήματα. Αυτό ε, είναι απαραίτητο. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα, δεν είναι εύκολο, αλλά τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. Το GSMR μετά, το, ραδιοσύστημα των uh, σιδηροδρόμων, ανήκει στο ETMS και με αυτό ασχολούμαστε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να συμπληρώσουμε την εκδοχή που λειτουργεί, που ισχύει και με την UIC πρέπει να κανονίσουμε ποια θα είναι τα μελλοντικά πρότυπα. Μία μικρή διακοπή εδώ. Συζητείται πολύ η δυνατότητα η υπηρεσία μας να έχει ένα ρόλο στην υποστήριξη της βιομηχανίας εκτός Ευρώπης. Σήμερα 50% των συμβάσεων για το ETMS και πάνω 50% το GSMR είναι με φορείς εκτός Ευρώπης. Έχουμε πολλούς εταίρους, καθορίζουμε προδιαγραφές που, για τη χρήση, έχουμε πολλές επαφές Βραζιλία ας πούμε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τώρα και από τις Ηνωμένε Πολιτείες κατέθεσε ένα αίτημα χτες. Άλλο θέμα αφορούσε το ρόλο της υπηρεσίας στην περίφημη του, περίπτωση του, του, της σύραγγας της μάχης, διότι επανειλημμένα αναφέρθηκε αυτό, η αποδοχή αυτών των σειρμών είναι θέμα των εθνικών φορέων ασφαλείας για την διόρυγα της μάχης υπάρχει ειδική υπηρεσία ασφαλείας που παίζει το ρόλο της και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών μελών που αναμειγνύονται στο όλο θέμα. Επίσης, καθορίσαμε ένα TSI για την ασφάλεια στο, στη σιδηροδρομική σύραγγα που βασικές αρχές είναι σχετικά απλές δεν υπάρχει περισσότερο βάρος για την ε, αμαξοστοιχεία και το σειρμό, αλλά κυρίως εστιαζόμαστε στις υποδομές. Αλλά υπάρχει μία εξαίρεση για τη σύραγγα, διότι για την ώρα δεν εμπίπτει στο πεδίο του TSI του συγκεκριμένου. Απ' την άλλη, ε, ξέρετε ότι η διμερή συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασίλειου ήταν ή είναι, δεν ξέρω τι να πω σήμερα, τροποποιήθηκε τέλο πάντων ή τροποποιείται και αυτή η διαδικασία συμπίπτει και με την προμήθεια των νέων, των νέων σειρμών από τη Eurostar. Σημειώσαμε, παρόλο που έγιναν κάποιες δηλώσεις στον τύπο ε, και υπάρχαμε πολλά τηλεφωνήματα από τους δημοσιογράφους, δεν μας ρώτησαν μέχρι τώρα να κάνουμε, δεν μας ζήτησαν να κάνουμε μια μελέτη, να ετοιμάσουμε τεχνική γνωμοδότηση ή να αναλύσουμε τη συμβατότητα των νέων κανόνων που προτείνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι τόσο φύς ε, η νομική βάση αν μπορούν και εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Ε, θα θέλαμε να αναθεωρήσουμε εν πάση περιπτώσει το TSI όσον αφορά την ασφάλεια στη σύραγγα της μάχης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσει για τις αμαξοστοιχίες για τη σύραγγα αυτή και θα ξεκινήσουμε τις εργασίες το 2011. Η όλη προβληματική θα καλυφθεί. Για την ώρα όμως δεν έχουμε επίσημο αίτημα να γνωμοδοτήσουμε επιτεχνικών θεμάτων για το συγκεκριμένο θέμα. Κάτι άλλο. Για το 2011 θα εστιαστούμε για την ασφάλεια, την αξιολόγηση του κινδύνου, θα εστιαστούμε πάνω σε αυτά. Κάνουμε πολλά περίπλοκα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν πολλοί και καμιά φορά ότι και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Αλλά είμαστε πεπισμένοι τώρα ότι ό,τι κάνουμε στο τομέα της ασφάλειας βοηθάει στον τομέα της λειτουργικότητας και τούμπαλιν. Τονίζοντας λοιπόν, τονίζοντας την αξιολόγηση του κινδύνου, βοηθάμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι ασύμβατοι κανόνε πρακτική που ακολουθούνται. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε μια κοινή προσέγγιση και κοινή διαδικασία που να ακολουθείτε. Είναι ουσιαστικό. Θέλουμε τα TSI να καλύπτουν όλο το συνδρομικό δίκτυο. Θέλουμε αυτό να γίνει μέχρι το 2012. Κάνουμε κάποιε προσθέσει στο ERTMS. Έχουμε νέε βασικέ γραμμέ για τι ραδιοσυχνότητες κλπ και μόνιμη προτεραιότητα είναι η συμβατότητα με παλιά συστήματα όσον αφορά τι επενδύσει και γενική αποδοχή. Έχουμε πολλού κανόνε για τη συνοριακή αποδοχή. Πρέπει να διευρύνουμε τη διαφάνεια τη προσβάσεω στα δίκτυα. Αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητα και βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουμε τη σταδιακή βελτίωση και εναρμόνιση στου τομεί αυτού. Και στον οικονομικό τομέα έχουμε όλο και περισσότερα αιτήματα να κάνουμε αξιολογήσει εκ των υστέρων και αυτό είναι σημαντικό. Συμπέρασμα λοιπόν. Αναπτύσσουμε πολλές δραστηριότητε. Ε, είμαστε σε επαφή, ε, μάλλον είμαστε σε επαφή με όλους τους στόχους, τους πετυχαίνουμε τους στόχους, δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλές απροσδόκητες αιτήσει που πρέπει όμως να συμμορφωθούμε, προέρχονται από τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές αρχές ασφαλείας, και από τον τομέα γενικά να ετοιμάζουμε κατάρτιση, ενημέρωση, διάδοση πληροφοριών διότι είναι γιγαντίο το πρόγραμμα τώρα. Είναι εύκολο να αποφασίσει στι Βρυξέλλες και αλλού κάτι, ότι θα έχουμε δύο συστήματα στην Ευρώπη για το πίσω μέρο των ε, σειρμών κλπ. Αλλά για να εφαρμοστεί αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουμε πολλέ αλλαγέ που πρέπει να κάνουμε σε φυστάμενου κανόνε και έχουμε προτεραιότητα από του χρόνου να κάνουμε την ε, απλούστευση. Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα που θα προσπαθήσουμε, κάτι που δεν είναι ποτέ εύκολο, ε, να τα κάνουμε πιο απλά. Και όταν έλεγα η διάδοση πληροφοριών δεν σημαντικό μόνο να έχουμε κοινού κανόνε, αλλά κοινή ερμηνεία, κοινή αντίληψη των κανόνων, κοινέ διαδικασίε για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Τέλο. Πιθανότατα είμαστε εμεί η υπηρεσία που ελέγχεται περισσότερο από όλε τι υπηρεσίε του τομέα των μεταφορών, από του εμπλεκομένου, από τα κράτη-μέλη, από την Επιτροπή Ρίσκα. Ε, βλέπω ότι παράγεται πάρα πολύ εργοκή. Η υπόλοιπη συνεδρία ΡΙΣΚ θα εξετάσει περίπου 50 προτάσεις. Το θέμα είναι πώς μπορούμε ίσως στο μέλλον να τα χειριστούμε καλύτερα τα πράγματα και συναντηθήκαμε εκπροσώπου του τομέα πρόσφατα και μα ζητά ο τομέα να επιταχύνουμε τι διαδικασίε. Όταν θα πάρουμε απόφαση, αν χρειάζεται, χρειάζεται μήνε για να μεταφραστεί κλπ. Και, και ίσω υπάρχει ένα περιθώριο ε, αν ρυθμιστεί αυτό να έχει περισσότερη ελευθερία φορέα. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Βισλέ. Ξεκινήσουμε με τα μέλη λοιπόν. Ο κύριος Σασάντα έχει το λόγο πρώτος. Dziękuję bardzo. Ja mam pięć pytań. Po tragicznym wypadku pociągu to... Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Μετά από το τραγικό ατύχημα του Βιαρέτζο στην Ιταλία του 2009, η ΕΡΑ έλαβε διάφορες αποφάσεις για την αύξηση της ασφαλείας, κυρίως όσον αφορά τα τρένα που μεταφέρουν εμπορεύματα αλλά δεν είναι απόλυτα σαφής για μένα αυτή η διαδικασία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για να αυξηθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων γενικότερα στην Ευρώπη. Δεύτερη ερώτηση. Ο ρόλος της υπηρεσίας σας συνίσταται στο να ε, έχετε πάρα πολύ σαφείς ε, αδειοδοτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφαλήτα. Προς το παρόν υπάρχουν για τα διάφορα κράτη διαφορετικές απαιτήσεις, πρέπει να γίνεται επαλήθευση ανάλογα με τα έργα υποδομής της κάθε χώρας και μετά από την αδειοδότηση θα έπρεπε οι σειρμοί να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν τα κράτη-μέλη απαιτούν αυτοί οι οποίοι ζητούν αυτή την αδειοδότηση να πληρούν και άλλα κριτήρια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Τι κάνει τι θα κάνει μάλλον η υπηρεσία σας στο μέλλον όσον αφορά αυτή την όλη διαδικασία αδειοδότησης των ε, σειρμών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Τρίτη παρατήρηση. Πρέπει επίσης εσείς να έχετε, για να μπορείτε να εξασφαλίσετε την διαλειτουργικότητα, μία σειρά τεχνικών προδιαγραφών να ισχύουν Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Οι τέσσερι που έχουν ε, υιοθετηθεί μέχρι τώρα δεν ε, επιλύουν το πρόβλημα, διότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών. Τα θέματα λοιπόν τα οποία ακόμη δεν έχουν καλυφθεί από το TSE καλύπτονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για κάθε χώρα και είναι ανοιχτά σημεία ακόμη, εκκρεμή. Εσείς θέλετε τώρα να, να ασχοληθείτε με αυτά τα εκκρεμή θέματα για να τα επιλύσετε. Αυτά λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία για τα open points όπως λέγονται, για αυτά τα εκκρεμή, τα θέματα ανοιχτά σημεία, είναι ακόμη χρονοβόρος. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει ακόμη να επιληθούν. Πού βρίσκεστε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία και πώς θα επιλύσετε αυτό το πρόβλημα των ανοιχτών σημείων σχέση με το RTMS. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει τάση να παρέμβει κανείς όλο και περισσότερο στο σύστημα των σιδηροδρόμων. Υπάρχει συντονισμός των προγραμμάτων ασφαλείας, Φερρυπίν. Δεν ξέρουμε όμως εσείς τι προτίθεστε να κάνετε. Στο μέλλον θέλετε εσείς να είστε πραγματικά ο ρυθμιστής αυτής της ενιαίας αγοράς των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν. Πρώτα απ' όλα, το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ζασάντα έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα και εγώ θα ήθελα να μάθω αυτά τα τελευταία έξι χρόνια πώς ε, στοχοθετήθηκε από στρατηγικής άποψης η ε, εργασία της ε, Ένωσης Σιδηροδρομών. Έχουμε θέσει 12 βασικά σημεία με 114 ε, συνεργάτες και αν τα δούμε αυτά στα πλαίσια και των ε, διορθωτικών ταμείων μπορώ να καταλάβω πολλο είναι να, να, συγκεντρωθούν, να συντονιστούν 27 κράτη-μέλη και να απαντήσουν ε, με βάση και τα εθνικά του συστήματα σιδηροδρόμων αλλά και με το γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο που έχει τεθεί. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις σε μία από τις μία τελευταίες μας συζητήσεις υπήρξε μία σαφής αναφορά ότι δηλαδή σε αυτό το τομέα πρέπει να εκπονηθεί ένας κατάλογος προτάσεων τον οποίο θα μας παρουσιάζεται για το πώς θέλετε να, ε, να, διαχειριστείτε αυτές τις απαιτήσει διαλειτουργικότητας που δηλαδή μπορούν να υπάρξουν, που υπάρχουν επικαλύψεις, που μπορούμε να συνδέσουμε τον ένα τομέα μεταφορών με τον άλλο. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία. Και αν δούμε, αν θέλουμε να κρίνουμε την, την κατάσταση του σύνολό τη, εγώ με λίγο, γιατί λέτε ότι τώρα έχουμε κάποιες ε, ρυθμίσεις για διαφόρους τομείς εργασίας για τα κράτη-μέλη, με, για, τα, για τους υδροδρόμους των κρατών μελών, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, για την ασφάλεια. Όλα αυτά θέλουμε να τα εξυλολογήσουμε, να δούμε πού υπάρχουν, ε, πού τέμνονται αυτές οι δραστηριότητες και αν υπάρχουν ε, ε, κοινά σημεία. Δεν μπορούμε απλώς να είμαστε επιχειρησιακοί. Τώρα μας είπατε ότι θέλουμε να εξοπλίσουμε τα, τα τρένα γιατί έχουμε πάρα πολλά τρένα τα οποία πρέπει να σταματήσουν να κινούνται. έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε μόλις 70.000 τρένα που να πρέπει να εξοπλίζονται τώρα είναι πολύ περισσότερα. Εσείς όμως ποιο είναι ο πυρήνας τώρα των εργασιών σας. Έχουμε τρία πακέτα για τους σιδηροδρόμους φέτος. Η Κομισιόν ε, αργά μεν, αλλά Εν πάση περιπτώσει ζήτησε από τα κράτη-μέλη αυτά που υπάρχουν στα τρία πακέτα για τους, ε, ε, για τους ε, για την έγκριση, των, για την μεταφορά και την ασφάλεια, την απελευθέρωση των, της κινητικότητας των αγαθών και των, και των ανθρώπων, να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και είμαστε τώρα στη φάση της αξιολόγησης. Εσείς Πώς εμπλέκεστε σε όλο αυτό, πώς ε, λαμβάνετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι σημαντικό σημείο αυτό. Στο μέλλον δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ε, προτεραιότητα που θα πρέπει να πάρουν τα αγαθά, να παίξουν ρόλο και οι ενιαίες θηρίδες. Γιατί υπάρχουν πολλές ε, υπηρεσίες στα κράτη-μέλη που ασχολούνται με τον ανταγωνισμό και θέλουν να απελευθερώσουν τον ανταγωνισμό θα είναι αυτό στα καθήκοντά σα ή θα πρέπει να υπάρξει δική μας ε, άλλο συντονισμό εν πάση περιπτώσει. Επίση, οι συνέργειες ναι είναι σημαντικέ, Με εκπλήσει όμως το ότι στην, για την απελευθέρωση του, των συνδρομικών μεταφορών διασυνοριακά μεταξύ Γαλλίας ας πούμε και Ηνωμένου Βασιλείου το θέμα της μάχης παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ε, καταρχήν δεν πρέπει να αλλάξουν οι εθνικές συμβάσεις έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να βρούμε συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Πώς θα δραστηριοποιηθείτε εκεί, πώς θα ηγηθείτε αυτού του τομέα έτσι ώστε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στα δίκτυα σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Και εγώ έχω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την ΕΡΑ. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ε, σιδηροδρόμων είναι 170 χρόνων στην ε, Ευρώπη. Και υπάρχει μεγάλος ε, μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, υπάρχουν συστήματα που δεν έχουν καλές συνδέσεις, τώρα έχουμε προβλήματα και διασυνοριακά τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και το πρόσφατο ε, δυστύχημα ε, στο Βέλγιο και αυτό ο τομέας της ασφάλειας είναι ο πιο σημαντικός επί του οποίου θα πρέπει να συνεργαστούμε. Νομίζω όμως ότι συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε ένα ενιαίο χώρο μεταφορών σιδηροδρομικών. Έχουμε και το πακέτο, για, το δεύτερο για τους, ε, για το οποίο ίδρυσε και τη δική σας υπηρεσία και ε, θήκες και της διαλειτουργικότητας. Δυστυχώς από αυτή τη θεωρία δεν έχει προκύψει καμία πράξη και διάφορα κράτη-μέλη παραπονούνται και το δικό μου βέβαια και άλλα για το ITCS και για αυτά που είπατε σήμερα να πω κάτι. Και για το σχέδιο της Λευκής Βίβλου αλλά και, για, και από, την, ε, από την ανακοίνωση της Κομισιόν ε, αναφέρεται ότι θα προκύπτει μάλλον ότι θα ενισχυθεί η ΕΡΑ ώστε να μπορεί να επηρεάζει όσο η ΕΜΣΑ και η EASA τα καθήκοντα της ΕΡΑ τα αναφέρατε και εσείς σε ό,τι αφορά την ε, εξισώση των, ε, ασφαλιών, των απαιτήσεων ασφαλείας στα κρατη την έγκριση, την δραστηριοποίηση κτλ, την πρόσβαση. Ε, και πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει εδώ ότι θα εξετάσει πώς θα μπορέσει να διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΕΡΑ. Και έρχομαι στο ερώτημά μου. Πρώτο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι αποτέλεσμα είχε αυτή η εξέταση, αυτή η μελέτη, πώς ε, σχεδιάζεται να ενισχύσετε περισσότερο την αέρα συγκεκριμένα. Δεύτερο ερώτημα προς την αέρα. Τι αρμοδιότητες θα θέλατε εσείς να έχετε ως υπηρεσία και πώς θεωρείτε ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τρίτο ερώτημα, πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μιλήσαμε και για, την, ε, για, το, για, την, για, τη σειρά της μάχης και το είπε και ο συνάδελφος Κουν. Εσείς θέλετε να έχετε εντολή να δραστηριοποιηθείτε στο τομέα αυτό ή θέλετε να ζητήσετε να γίνει μελέτη σε ό,τι αφορά την περαιτέρω δραστηριοποίηση, σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας. Ε, άλλο ερώτημα προς την ΕΡΑ. Σε ό,τι αφορά το, η βάση δεδομένων σας, γιατί ακούσαμε ότι δεν λειτουργεί πολύ καλά. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την εισαγωγή των ενιών θηρίδων. Ε, πόσο θα εμπλακείτε εσείς όλη αυτή τη διαδικασία, θα την εποπτεύσετε καθόλου. Και ένα τελευταίο ερώτημα πάλι προς την αέρα. Σε σχέση με το, ε, ενσωματωμένο, την ενσωματωμένη, ε, ε, ολοκληρωμένη μάλλον έκδοση εισιτηρίων. Αυτό γίνεται να εφαρμοστεί και στους σιδηροδρόμους. Αυτά, Πρόεδρε, τα συγκεκριμένα ερωτήματά μου από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, οπότε δεν άκουσα από την αρχή τις παρατηρήσεις. Διαπίστωσα όμως, ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση για δραστηριοποίηση στο μέλλον. Ο συνάδελφος Κιούν ανέφερε την θέση του ΕΛΚ, οπότε εγώ θα περιοριστώ απλώς σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και σε κάποια ερωτήματα. Πρώτον, να ρωτήσω κι εγώ αν εσείς ως πρόεδρος είσαστε της άποψης ότι η ΕΡΑ διαθέτει αρκετά επαρκή κονδύλια και αρμοδιότητες. Νομίζω ότι πολλοί κανόνες εμπίπτουν στις, εθνικές, ε, στις αρμοδιότητες των εθνικών ε, αρχών. Και επίσης διαπίστωσα ότι είναι, δεν, μπορούν, δεν έχουν τα κρατημέλη πάρα πολλούς ε, επαρκείς μάλλον πόρους και έχουν και πάρα πολλές αρμοδιότητες για να μπορέσουν να τις ε, ελέγξουν και να τις εποπτεύσουν ε, όπως ας πούμε οι απαιτήσει της εργασίας των εργαζομένων οι οποίες έπρεπε υποτίθεται να ρυθμιστούν από το 2005 εν τω μεταξύ, όμως οι συνθήκες εργασίας όπως είχαν συμβοληθεί δεν έχουν τηρηθεί. Οπότε εμείς ως ε, Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι οι συνθήκες εργασίας και οι σχετικές ε, ε, διατάξεις θα πρέπει να βελτιωθούν, ειδικά για τους οδηγούς των σειρμών. Προς το παρόν βλέπουμε μόνο επιδείνωση των συνθήκων εργασία τους. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες, πώς μπορούμε να, να υποπτεύσουμε και να ελέγξουμε ότι θα τηρούνται αυτέ οι συνθήκες. Τώρα, το ERTMS το οποίο ζητείται να είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμο. Ας πούμε μια μικρή χώρα. Για κάθε, για κάθε σειρμό υπάρχουν τρία-τέσσερα συστήματα ασφάλειας. Αν τώρα θέλουμε να, αν θέλει ένα σειρμός να, να ταξιδέψει διασυνοριακά, αυτό καταρχάς είναι μεγάλο ε, οικονομικό βάρος και δεύτερον είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι διαλειτουργικό, τα, να είναι διαλειτουργικό το σύστημα διασυνοριακά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ασφαλείας μέσω των διαφόρων ε, συστημάτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να πλουστεύσουμε τις διατάξεις και να, τα, ε, να διευκολύνουμε την κατάσταση. Το ζητούν και τα κράτη-μέλη. Μετά, ο συνάδελφος Έρτοκ το είπε, αυτό με την βάση δεδομένων. Μου είπαν και εμένα ότι η οι απαιτήσει αυτέ, οι προποθέσει για τη χρήση των σιδηροδρόμων δεν, ε, είναι επαρκώς, δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς στη βάση δεδομένων. Αν ας πούμε κάποιος θέλει να κάνει να έχει τέτοιε δραστηριότητε διασυνοριακά, είναι πολύ δύσκολο να βρει τι προποθέσει που πρέπει να τηρήσει για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί. Ε, αν θέλει ειδικά να, να έχει δραστηριότητε τέτοιε διασυνοριακά μέσα σε τρία-τέσσερα ε, κράτη-μέλη. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούγκια. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει σύντομε έχω. Η πρώτη αφορά τα συνδρομικά ατυχήματα. Διότι πέρα από τα φετινά ατυχήματα. Θα ήθελα να ξέρουμε ενημέρωση από την Έρωση να αφορά τα ατυχήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, όπως αυτό του Βιαρέτζο. Το Βιαρέτζο τραγικός είναι ένα παράδειγμα συντονισμού ευθυνών, διότι υπάρχει μια ευθύνη ενδεχομένως από πλευράς του χειριστού του δικτύου, ενδεχομένως ευθύνη του ιδιοκτήτη του τρένου, ενδεχόμενη ευθύνη και των συντηρητών εσείς θα πρέπει να παίξετε πιο αποφασιστικό ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρετε αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πιο πρόσφατες ε, πληροφορίες για τις έρευνες που διεξάγονται φέτος. Συμμετείχατε στο σεμινάριό μας όσον αφορά την ασφάλεια, κάνοντας και μια ομιλία λαμπρή που την εκτιμήσαμε. Θα ήθελα να ξέραμε αν μπορείτε να μας δώσετε πιο πρόσφατες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον προπολογισμό ε, ε, του οργανισμού. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την απαλλαγή εκ μέρους της Επιτροπής και είδα ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, ανέφερε την καθυστέρηση όσον αφορά την απορρόφηση, τη χρήση των πόρων που διαθέσαν την υπηρεσία και τη διοργάνωση των διαγωνισμών για τις προμήθειες. Ήθελα να ξέρω κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό και πάνω σε αυτό αν υιοθετήθηκαν καλύτερες διαδικασίες για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βισλάιπη, και εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Χέρτσογκ. Δηλαδή, βάσει δεδομένων, τη βάση δεδομένων γεωράτης Έχω στενούς δεσμούς με κάποια από τα πανεπιστήμια, το Newcastle, το Manchester, ακόμα και με την Καλσρούη, το τεχνικό πανεπιστήμιο, τεχνικά πανεπιστήμια που τα επεξεργάζονται και εκφράζονται ανησυχίε από τα πανεπιστήμια ότι βάσει δεδομένων γιουράτη δεν δουλεύει, α το πούμε έτσι. Και έχει και ένα και προβλήματα. Ένα παράδειγμα μου έδωσαν. Αν ψάξει, α πούμε, εκτροχιασμοί για όλες τις χώρες των εμπορικών τρένων σου δείχνει 17 εκτροχιασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν κάνεις το ίδιο ψάξιμο για το Ηνωμένο Βασίλειο στο δικό σας σύστημα δείχνει άλλο στοιχείο, άλλο αριθμό βγάζει με την έρευνα. Και διατείνονται ότι είχε, το πρόβλημα είναι ότι το, το Eurostat και το Euratis, τα δύο συστήματα, και το ερώτημα είναι γιατί να μην έχουμε μία νέα βάση δεδομένων που λειτουργεί σωστά. Ένα κωδικοποιημένο σύστημα παρόμοιο με των Αμερικανών και των Καναδών. Σας το θέτω λοιπόν. Πρώτα αυτό, δεύτερο. Άλλο θέμα που έθεσαν οι πανεπιστημιακοί. Ε, υπάρχει ένας διαγωνισμός για μία μελέτη για τους εκτροχιασμούς. Ποιος είναι ο ανάδοχος, ξέρουμε και αν ξέρουμε. Είναι ικανοί όσον αφορά τα θέματα αυτά. Έχουν τις γνώσεις τις ιδεοδρομικές, οι ανάδοχοι. Και το τελευταίο. Εσείς σαν ERA, σαν ΕΡΑ, πώς έχετε σε επαφή με τους ερευνητικούς φορείς και τα πανεπιστήμια. Και τα πανεπιστήμια λοιπόν για την έρευνα και τα όσα συμβαίνουν στο σιδηροδρομικό τομέα και κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Όπως θα είδατε, αυτό είναι κάτι που ασχολεί ιδιαίτερα τα μέλη, κυρίως μετά από πρόσφατα ατυχήματα. Χαίρομαι που αναφέρθηκε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των φαναριών των τρένων στο τέλος των σειρμών, και από ένα μικρό σπόρο μεγαλών μεγάλα δέντρα, δηλαδή έχουμε το σπόρο, έχουμε το κουκουνάρι, αν θέλετε το βελανίδι, που είναι τα φώτα του τέλους του σειρμού και επίσης τι άλλα προβλήματα θα λύσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά οι σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές είναι άλλο θέμα. και με τους υπευθύνους των σιδηροδρόμων των κρατών μελών. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στους σιδηροδρόμους της Ευρώπης όσον αφορά τις εισφορές για τις υποδομές και τα διάφορα συστήματα για την επιβολή τελών για τη χρήση των ε, υποδομών. Για τη σύραγγα ε, της μάχης έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Wembley μέχρι το σύραγγα ένα σύστημα, μέσω από, το, από τη σύραγγα δεύτερο σύστημα, από τη σύραγγα στη Γαλλία τρίτο σύστημα. Είναι αποδοτικό αυτό. Αυτό πώς θα προωθήσει καλύτερη χρήση των σιδηροδρόμων στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες όσον αφορά τη σύραγγα της μάχης. Πώς να το πω τώρα. Έχει ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις, τους κανόνες, τις ρυθμίσεις και ε, τις ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια. Να σας πω σαν Βρετανός κάτι. Δεν θέλω να στενοχωρήσω κάποιους από τους Γάλλους συναδέλφους λέγοντας αυτό. Σαν Βρετανός λοιπόν, σκασίλα μου ποιος φτιάχνει το τρένο. Από τη στιγμή που το τρένο είναι ασφαλές, γρήγορο, αποτελεσματικό και κάνει τη δουλειά για την οποία σχεδιάστηκε και από τη στιγμή που μεταφέρει τον κόσμο και τον περνάει από τη σύραγγα γρήγορα. Δεν μπορώ να κολλήσω εδώ πέρα. Πρέπει να είναι τόσο μήκο μετά άλλο μήκο και αυτό ο παντογράφο, ο άλλο παντογράφο, αυτή η πρόσβαση, την άλλη πρέπει να έχει. Θέλω ένα τρένο να περάσω από τη σύραγγα. Αυτό είναι όλο. Αυτά και ευχαριστώ. Θέλει η Κομισιόν το λόγο ή θέλετε να περιμένετε. Μετά τον ε, κύριο Βέσλαϊ. Πολύ έξυπνο. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω και στα γαλλικά. Euh, λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, η ασφάλεια, το Βιαρέτζο και τι έγινε. Πολλά θέματα λοιπόν όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε κοινού δείκτε και κοινέ μεθόδου για να μπορέσουμε να έχουμε συγκρίσιμε ε, αναλύσεις. Νομίζω ότι οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες και στο ίντερνετ, πρέπει να τις μελετήσετε, θα είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην περίπτωση του Βιαρέτζο, που ήταν ιδιαίτερα δραματική περίπτωση, και στην περίπτωση του ατυχήματο του Μπούζιγκεν στο Βέλγιο, που είναι τα πιο εντυπωσιακά και γνωστά ατυχήματα, θα πω το εξή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και θα πρέπει να διαβάζετε τι εκθέσει που κάνουμε εμεί για την ασφάλεια. Λοιπόν, δύσκολο να το πούμε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων όλο και επιβελτιώνεται. Πέρσι είχαμε θύματα. Παρά το ατύχημα του Βιαρέτζο, μικρό αριθμό αν θέλετε και τώρα σε επίπεδο Ευρώπης το επίπεδο ασφαλείας Έχουμε 40 με 50 θανάτους ε, ετησίως, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γύρω στους 300. Και σε σχέση με τα ε, τροχαία ατυχήματα καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Αλλά βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Μετά από το ατύχημα του Βιαρέτζο, ο κύριος Ταγιάννη οργάνωσε μια διάσκεψη και μαζί με όλους τους ειδικού εξετάσαμε όλα τα τεχνικά μέσα, επιμένω, για την ασφάλεια των σειρμών για τις επικίνδυνες ουσίες, τα επικίνδυνα υλικά και ήδη υπάρχουν γύρω στα 20 μικρά τεχνικά μέτρα τα οποία παρά το γεγονός ότι λέγονται μικρά και επηρεάζουν θετικά και την ασφάλεια. Παρά τις έρευνες που έγιναν, πρέπει να πω ότι δεν έχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι ε, των ε, Βελγικών Υπουργείων εμπλάκημεν από την πρώτη μέρα που έγινε το ατύχημα στο Μπούζιγκεν. Τώρα, η δικαστική έρευνα, η αστυνομική συγγνώμη, έρευνα ε, στην Ιταλία έγινε και εκείνοι έχουν αναλάβει την όλη έρευνα. Έχουμε εμεί κάποια στοιχεία από τους υπεύθυνου ε, της Ιταλίας, αλλά ίσως υπάρχει και θέμα νομικό στη μέση. Τώρα, το πρόβλημα των διαφορετικών STIs, αυτά τα open points που αναφέρεται μεταξύ των ε, διαφόρων κρατών μελών. Όλα τα θέματα που δεν μπορούν επί δεκαετίες να επιλύσουν οι ειδικοί επισυροδρόμων είναι αυτά τα περίφημα open points. Και όντως υπάρχουν πολλά θέματα. Ακούστε, υπάρχει ε, Εγώ όταν γίνονται επικρίσεις ε, για τους σιδηροδρόμους λέγω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάποιοι άλλοι δείκτες έχουμε διάφορες γραφικές ε, παραστάσεις που μας δείχνουν την ε, πρόοδο, την ασφάλεια το θέμα της τροχοπέδησης, των ε, σειρμών. Το τέλμες είναι ένα θέμα το οποίο το μελετάμε και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι επιταχύνουμε το ρυθμό της εργασίας μας. Είναι όμως σαφές ότι η επίλυση των open points όντως είναι η πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη διετία των μονάδων που ασχολούνται με τη διαλειτουργικότητα. Τα RTMS, για να κάνω μία μικρή ιστορική αναδρομή. Πρέπει να σας πω ότι είναι το μόνο και ίσως, το πρώτο και ίσως το μόνο καθήκον για το οποίο εμείς έχουμε μια κάποια εξουσία. Έπεσε σε εμά αυτή η ευθύνη. Η μικρή μας ομάδα που αποτελεί την εποχή του μέσα από δύο άτομα, σε ένα χρόνο κατόρθωσε με τον κλάδο να θεσπίσει τον κανόνα 3.0D. Και είδαμε όταν ασχοληθήκαμε με το όλο θέμα ότι υπήρχαν προβλήματα. Πρέπει όμως να σας πω ότι με τις πολύ μικρές ομάδες δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα συμμόρφωσης. Δεύτερον, ένα άλλο αποκαλυπτικό στοιχείο. Όταν τέθηκε σε ισχύ το σύστημα αυτό, αυτό που άλλαξε σε σχέση με το παρελθόν ήταν ότι η υπηρεσία μας έκανε το Change Control Management, την διαχείριση του συστήματος ελέγχου για την αλλαγή του RTMS. Και πρέπει να σας πω ότι συνέβη αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν υπάρχει πιλότος στο αεροπλάνο, δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να ηγηθεί όλων των αλλαγών που έπρεπε να γίνουν. Είναι ε, λοιπόν η δουλειά που έγινε τρομερή. Είμαστε δύο, τώρα είμαστε δώδεκα στην ομάδα αυτή. Όλοι θέλουν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα αυτό να προχωρήσουν τα πράγματα και όλοι προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση, άρα έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Και βεβαίως συνεχίζουμε να κάνουμε τις βελτιώσεις και τις αλλαγές στο παρόν σύστημα, πράγμα που το επιτρέπει να λειτουργεί. Και αν θέλω να σας πω ότι σήμερα το RTMS αφορά ένα ε, σύστημα που το RTMS ισχύει για τις μισές χώρες της Ευρώπης, πρέπει να σας πω ότι καλύτερα να πάρουμε από το ράφι ένα καινούριο σύστημα και το εφαρμόσουμε σε όλους, παρά να προσπαθήσουμε να κάνουμε διορθώσεις για να ισχύσει ένα σύστημα διαφορετικό για όλους μετά. Τώρα, ο συντονισμός των αρχών ασφαλείας ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Είναι ένα θέμα το οποίο υποτιμούν κάποιοι, ήταν όμως το πρώτο καθήκον μας. Καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικές ε, ε, δυσκολίες εκ μέρους κρατών μελών, διότι πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κράτη ε, που δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι από κοινού να βοηθήσουμε τους πάντες και έχουμε πραγματικά ε, πολλά αιτήματα ε, για να βοηθήσουμε τέτοιου είδους αρχές να δημιουργηθούν. Δώσω το παράδειγμα της ε, Σλοβενίας, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά σε τρία χρόνια, αλλά ακόμη υπολείπονται πολλά. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε εμείς να συντονίσουμε όλες τις εθνικές αυτές αρχές, να θυσμίσουμε τις εθνικές αρχές για να συντονιστούν τα θέματα. Πολλές ερωτήσεις για ενδιαφέρουσες έκανε ο κύριος Κούν. Πρώτα απ' όλα είναι προφανές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία σε αυτό το μοσαϊκό που διαφορετικών συστημάτων στους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη. Εγώ εργάζομαι εδώ, εδώ και τέσσερα χρόνια και αρχίζω και το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι θεμελιώδους σημασίας. Όλη η δουλειά που έγινε στα πλαίσια της αμοιβαία αποδοχής είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας χιλιάδες διαφορετικούς κανόνες. Με το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα ε, θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, διότι στο παρελθόν ρωτούσαμε γιατί ισχύει ο κανόνα και μα λέει μη σα νοιάζει, έτσι εφαρμόζεται, δεν μπορούμε να σα πούμε τίποτα άλλο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη αμοιβαία αποδοχή θα χτενίσουμε το όλο σύστημα και θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε κοινέ προδιαγραφέ. Ποια είναι η δυσκολία. Πολλά πράγματα τα οποία σήμερα κάποιοι μας ε, αρνούνται να μας αποκαλύψουν είναι κάποιες ε, πρακτικές ε, πολλές φορές υποχθόνιες για τις οποίες δεν υπάρχει διαφάνεια. Εμείς θέλουμε διαφάνεια και αιτιολόγηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως τώρα δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ότι αναθεωρημένη οδηγία για την διαλειτουργικότητα ισχύει. Όταν λοιπόν μια Εθνική Αρχή Ασφαλείας εγκρίνει ότι είναι σύμφωνο με το LTC, δεν πρέπει να αρχίσει και δεν μπορεί να αρχίσει ε, να εφαρμόζει μη διαφανείς εθνικούς ε, κανόνες και κανονισμούς. Αν υπάρχει παραμικρή υπόνοια θα πρέπει κανείς να προσφύγει κατά της χώρας αυτής στην Κομισιό. Υπάρχουν τα μέσα τα οποία μας το επιτρέπουν. Αρχίζει, αρχίζει. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα τομέα στον οποίο το πνεύμα φιλίας ήταν μια αρετή που πολύ διέθεταν στο παρελθόν. Η... Τώρα, οι κανόνες, ε, οι λειτουργικότητες και οι επιχειρησιακοί κανόνε πρέπει να θεσπιστούν από όλου για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την παραγωγικότητα. Τώρα, το θέμα της σύραγγας της μάχης Ήμουν απόλυτα σαφή. Η υπηρεσία μας δεν έχει καμία εξουσία, παρά μόνο για το RTMS. Αν μας ζητήσουν κάτι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι εύκολο, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι εθνικές αρχές και κυρίως η αρχή της σύραγγας που έχει την ευθύνη. Προσπαθώ να συνοψίσω, λέει ο μιλητής ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βάσει δεδομένων, πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλέ, ίσω υπερβολικά πολλέ. Προσπαθούμε λοιπόν, επειδή αναφέρονται τα μέσα, να σχεδιάζουμε την πολιτική μας. Αρχίσαμε με δύο άτομα και εδώ και πέντε χρόνια τρέχουμε πίσω από τα καθήκοντα που έχουμε. Και πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Στα θέματα πληροφορικής έχουμε 14 15 καθήκοντα σε θέματα πληροφορικής που χειρίζονται αυτή τη στιγμή 6 άτομα. Και όταν αναφέρεται η καθυστέρηση για τις ε, κρατικές προμήθειες, τις δημοσιοφορίες, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε την, την ε, προκήρυξη ε... για να ενισχύσουμε το όλο σύστημά μας. Πρέπει όμως να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Τώρα, Έχουμε, είπα, διαφορετικές βάσεις δεδομένων που είναι εικονικά δίκτυα στα οποία υπάρχουν τα στοιχεία που μας δίδουν τα κράτη-μέλη. Εμείς τα συμπληρώνουμε, αλλά εμείς καταρχήν εμπνεόμαστε από τα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Και δε, βεβαίως δεν λέγω ότι είμαστε τέλειοι και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι πρώτα απ' όλα να παρέχουμε στοιχεία μέσω της βάσης δεδομένων μας στην βιομηχανία του κλάδου, στις αεροδρομικές εταιρείε, αν θέλετε. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή σας για την σχέση μας με την έρευνα και τους ακαδημαϊκούς ε, κύκλους. Όντως είπαμε ότι εμείς θα πρέπει να παίξουμε συντονιστικό ρόλο πιο σημαντικό το κάνουμε ετήσι κάποιου, δεν είναι στα πλαίσια των κανονικών μας καθηκόντων. Όταν οι γενικές διευθύνσεις Φερρυπίν μας ζητούν να συμμετάσχουμε σε μία αξιολόγηση, το κάνουμε, αλλά είναι μία περιθωριακή ε, απασχόληση. Η ενιαία φυρίδα. Ο στόχος είναι πολύ απλός. Θέλουμε να το καταστήσουμε αυτό δυνατόν. Τι σημαίνει. Δηλαδή, εναρμονίζοντας τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, θα έχουμε την, δικα... την ε, δυνατότητα να εισαγάγουμε στο σύστημα την έννοια Προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε το μέσον που θα επιτρέψει να υπάρξει αυτό και οι υπεύθυνοι της εμπορίας, της αγοράς θα το εφαρμόσουν. Ο κύριος Μπάκαν έφερε τις αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες μας είναι πολλαπλές, αλλά δεν έχουμε εξουσία όπως σας είπα. Όσον αφορά τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας, κυρίως για τους οδηγούς, προχωρούμε για την ε, πιστοποίηση των κέντρων κατάρτισης και εδώ, όπως και σε άλλους τομείς, αλλά ακόμη αυτό δεν είναι στα άμεσα καθήκοντά μας, όλα εξαρτώνται και από τον ε, έλεγχο που θα υπάρχει στα εθνικά κέντρα πιστοποίησης. Σε θέματα ασφαλείας πρέπει να πω ότι επίσης έχουμε προχωρήσει πολύ προς το παρόν και τον έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας. Αναφέρθηκε ο προϋπολογισμός και εδώ σας αναφέρω δύο προβλήματα. Ο προ, είναι αυτό που είναι. Είπαμε ευθύ εξ αρχή ότι ο τίτλο 1 και 2 είναι ανεπαρκή και ο τίτλο 3, δεν το θέλω να το πω εδώ στο κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να σα πω ότι θα μα ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέσα του τίτλου 3, διότι η πραγματομοσύνη βρίσκεται εδώ. Και όντω, όταν γίνεται λόγο για τι ε, ε, κρατικές προμήθειες, θα θέλαμε τα πράγματα να τα κάνουμε εμείς όπως μπορούσαμε πολλές φορές χρησιμοποιούμε άλλους πόρους. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι πολλές φορές καθυστερούν όλες αυτές οι διαδικασίε των προμηθειών και δεν θα σα εκπλήξω λέγοντά σα ότι οι κοινοτικέ διαδικασίες είναι πραγματικά χρονοβόρες. Ραντί και Eurostat. Συνεργαζόμαστε με τη Eurostat. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν άλλα σημεία τα οποία αναθέτηκαν. Τώρα, για την ε, ρόλο των ρυθμιστών και για τα ε, τέρια, το ποιον βαρύνουν. Δεν έχουμε ε, εμείς σχέση με τους αυτούς οι οποίοι κάνουν τις ρυθμίσεις. Δυστυχώς προς το παρόν λοιπόν δεν ασχολούμεθα Δύο τελευταία στοιχεία. Περισσότερη εξουσία στην υπηρεσία μας. Το μέλλον μας θα αποφασίζεται από τις αρχές. Εμείς δεν έχουμε λόγο. Έχουμε ε, κάποια σχέδια, τα ολοκληρώνουμε, συζητούμε την Επιτροπή, με τους διάφορους φορείς, με τους εμπλεκόμενους και όλοι μαζί ελπίζω ότι θα συνεισφέρουμε στο μέλλον και στην τις υπηρεσίες αξιολόγηση για το μέλλον. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε. Έκανα μία ερώτηση για το αν έχετε, κάνει την, έχετε αναθέσει τη μελέτη για τους εκτροχιασμούς προς το παρόν. Όχι. Λοιπόν, ο κύριος Γκρίλο έχει 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αξιολόγηση της υπηρεσίας. Σημεριζόμαστε πλήρως την ανάλυση του κύριου Φερσλίπ για τα έργα που έγιναν κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ύπαρξής της. Δηλαδή, ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες μας η υπηρεσία. Προσδοκίες που είχαμε όταν είπαμε ότι πρέπει να συσταθεί. Στον τομέα της διαλειτουργικότητας, οι εργασίες υπηρεσίας ε, πέτρεψαν να υιοθετηθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις για την λειτουργικότητα όσον αφορά την ασφάλεια, η υπηρεσία. Ανέπτυξε κοινή προσέγγιση σε θέματα ασφαλείας, δηλαδή έχουμε τώρα εναρμονισμένους ορισμούς σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τους δίκτες ασφαλείας, έχουμε κοινούς στόχους ασφαλείας, μια πρώτη σειρά, την οποία βεβαίως θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω και έχουμε και τις κοινέ μεθόδους ασφαλείας, κυρίως την μέθοδο που αφορά την ανάλυση κινδύνων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για την πιστοποίηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά το RTMS, όπως ξέρετε έχουμε μία ε, σταθερή εκδοχή που χρησιμοποιούνται σε όλους τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ανά την Ευρώπη και όσον αφορά την ε, αμοιβαία αποδοχή για το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιεί. Η θέση των κρατών μελών είναι θετική σε σχέση με τα μέσα που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ όλων των κανόνων και να ε, πιστοποιείται η ισοδυναμία. Όσον αφορά το μέλλον, όπως είπε και ο κύριος Φερσλίπ, αυτή τη στιγμή γίνεται αξιολόγηση εξ έτσι όπως το προβλέπει ο κανονισμός. Και τα αποτελέσματα θα έχουμε του χρόνου το Μάρτιο. Στις 10 Δεκεμβρίου ήδη θα γίνει ένα σεμινάριο με όλους τους ενδιαφερομένους, με μια πρώτη εκδοχή αυτής της και πρώτη παρουσίαση αυτής της αξιολόγησης. Όσον αφορά τα πέντε επόμενα χρόνια και τις προτεραιότητες, Βεβαίως πρέπει να θέσουμε και προτεραιότητες. Για την διαλειτουργικότητα η προτεραιότητα είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών, διότι αφορά μόνο το ευρωπαϊκό δίκτυο και θα πρέπει να επεκταθούμε περαιτέρω στο σύνολο του συνδρομικού δικτύου όσον αφορά την ασφάλεια. Ήδη την αναφέραμε εδώ. Πώς πρέπει να ενεργήσουμε, ώστε όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό ατύχημα, όπως αυτό το Βιαρέτζο, να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Προσπαθούμε λοιπόν να θεσπίσουμε, να δημιουργήσουμε μία ομάδα εργασίας, η οποία θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ τα θέματα αυτά ασφαλής και θα πάρει τις ε, κατάλληλες απαιτήσεις όσον αφορά το RTMS. Έχουμε την εκδοχή 3, η οποία αυτή τη στιγμή μελετάτε για να μπορέσει να τελειοποιηθεί και να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά την αμοιβαία αποδοχή των σειρμών, θα πρέπει να έχουμε ένα πίνακα εύκολο που να μπορούν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιούν για να ξέρουν ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν και να είναι κοινώ αποδεκτοί ανά την Ευρώπη. Τώρα, Γίνεται λόγος για την ενίσχυση του ρόλου της υπηρεσίας. Όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα εργασία της 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού της Υπηρεσία και του χρόνου θα κάνει μια ανάλυση αντικτύπου και επιπτώσεων για να δοθεί πιο σημαντικός ρόλος στην υπηρεσία. Είπαμε προς τα πού θα πρέπει να κατευθύνουμε την μελέτη αυτή ενισχυμένο συντονιστικός ρόλος, ρόλος εποπτείας των εθνικών αρχών ασφαλείας, δεδομένου ότι οι έρευνες αποδεικνύουν ότι σε πολλές χώρες Φερρυπίν, οι εθνικές αρχές ασφαλείας δεν έχουν επαρκές προσωπικό για να φέρουν σε πέρας όλα τα καθήκοντα που τις έχουν ε, ανατεθεί σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. Μπορεί λοιπόν η υπηρεσία να τους βοηθήσει και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα αν χρειάζεται. Αυτό είναι ο πρώτος ρόλος, συντονιστικός και εποπτείας. Δεύτερον, όπως είπε ο κ. Φεσλίπ, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες κατάρτισης και διάδοσης των πληροφοριών είναι αρκετά εύκολο να υιοθετηθούν τεχνικές προδιαγραφές ή κοινέ μέθοδοι ασφαλείας. Θα πρέπει όμως να μπορούν και να εφαρμοστούν επιτόπου, στην πράξη. Πράγμα που ζητά να γίνει πολλή δουλειά σε επίπεδο κατάρτισης, ενημέρωσης πρώτα απ' όλα και κατάρτισης. Και επίσης υπάρχει το εξής θέμα η ίδια η υπηρεσία μπορεί να δίδει πιστοποιητικά θέσεις σε κυκλοφορία σειρμών ή πιστο, να το ικανό μιας ε, επιχείρησης. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε αρχίσει να συζητούμε για να δούμε κατά πόσο θα ήταν αποδοτικό να ζητήσουμε κάτι τέτοιο στην υπηρεσία, την οποία βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε και τα κατάλληλα συμπληρωματικά ε, κονδύλια. Άρα τίθεται εδώ και θέμα χρηματοδότησης και ύπαρξης κονδυλίων. Το, το Eurotunnel, η σύραγγα, μας απασχολεί το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι έγινε πριν από την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. Είναι λοιπόν φυσιολογικό να μην είναι, αν θέλετε, η σύραγγα ε, απολύτως ε, με τις διάφορες τεχνικές προδιαγραφές. Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς αναδρομικά να ζητήσει από κάποιον να πληρεί κάποια τεχνικά κριτήρια. Οι αρχές, οι υπεύθυνε μας έστειλαν τους, ε, τα σχετικά ε, τεχνικά θέματα. Τα είχαμε ζητήσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Πέρσι στα πλαίσια της ασφαλείας επίσης μας είχαν κοινοποιηθεί αυτοί οι κανόνες ασφαλείας. Και αυτή τη στιγμή με ανταλλαγή επιστολών με τις αρχές της σύραγγας εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αν μετά από την κοινοποίηση αυτών των κανόνων θέλει κανείς να κάνει κάποια αλλαγή θα πρέπει να τους κοινοποιήσει πρώτα στην Κομισιό για να δούμε εάν δεν υπάρχουν διακρίσεις και αν δούμε ότι μπορούν να υπάρχουν αρνητικές διακρίσεις μπορούμε να ζητήσουμε και τη συνδρομή της υπηρεσίας και ενδεχομένως να σταματήσουμε την εφαρμογή κάποιου κανόνα ο οποίος δεν θα είναι σύμφωνος με τα σημερινά κριτήρια. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε. Από τις διάφορες παρεμβάσεις κατάλαβα ότι υπάρχει για την ε, ταχύτητα των τεχνικών ε, προδιαγραφών μια κάποια δυσαρέσκεια. Έχουμε εκατομμύρια χιλιόμετρα, εκατομμύρια τροχαίο υλικό, σειρμούς. Πολλές φορές έχουμε σειρμούς 25 ετών παραπάνω, ε, σύραγγες 50-100 ε, ετών. Μην πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε αρμόνι σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 5 χρόνια λοιπόν. Γι' αυτό θέτουμε προτεραιότητες και μία από τις προτεραιότητες είναι αυτή η περίφημη διάδρομη για το ΦΡΕΤ για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να επιτύχουμε με την εγκατάσταση των συστημάτων RTMS την ε, ε, εναρμόνιση, την τεχνική σε μια πρώτη φάση πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα έχουμε πλήν εναρμόνιση πριν από πέντε χρόνια, αλλά θα το εκτιμούσα να το, δώσω πριν, να το δω πριν πεθάνω και αρχίζω να βάλω αν θα υλοποιηθεί αυτό και κατά τη διάρκεια ζωής των παιδιών μου. Εκτιμούμε τις δυσκολίες, τις τεχνικές και τα μέλη ήταν πολύ διπλωματικά, πρέπει να τα ακούσετε, όταν ο κύριος Λούντβικ θα έρθει από την CR. Α, θα το την Και είναι και καλός άνθρωπος, αλλά, αλλά υπάρχει αυτή η απογοήτευση, αυτή που από τα μέλη. Όσον αφορά τη σύραγγα τη ε, μάχη, συνεχίστε, συνεχίστε. Κύριε Έρθοκ, θέλετε να παρεύετε συντομία πριν αλλάξουμε τρόπο και πάμε στα κύματα και στους ωκεανούς με τον κύριο Ντερόιτερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εγώ είμαι απογοητευμένος ε, γιατί από τα ερωτήματα που έθεσα δεν απαντήθηκε κανένα. Εγώ ρώτησα ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε πριν από 1,5 χρόνο. Τίποτα δεν μου είπατε. Οπότε ε, σας ξαναλέω ότι εγώ απογοητεύτηκα πλήρως διότι δεν λάβαμε καμία, α, καμία πληροφορία από αυτά που είπε η Κομισιόν και θα ήθελα να καταγραφεί αυτό. Okay, may... Καλώς κύριε Χέρσογκ. Ίσως λοιπόν ο κύριος Φερσλέιπ αν έχει χρόνο να κοιτάξει τις σημειώσεις του και αν βρει αυτό που είπατε ίσως να αντιστοιχεί στις απαντήσεις. Λοιπόν, αν και οι δύο κυρίοι μπορείτε να δείτε αυτά που είπε και ο Σέτσοκ και αν κάτι χάσατε θα σας επαφήμαστε. Κύριε Βεσλάιπ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμούμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχετε, το ρόλο που έχετε και όπως σας είπα και το λέω σε όλους τους οργανισμούς, δεν είμαστε εδώ για να επικρίνουμε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε γιατί στο κάτω-κάτω αυτό που θέλουμε ε, είναι πολύ καλός οργανισμός Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και μαζί με τους άλλους οργανισμούς να δίνει τις μεταφορές που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ εκ νέου. We go from swaying carriages to swaying ships, if Mr. De Πάμε λοιπόν στα πλοία. Ο κ. Ντερόιτερ, κάπου εδώ είναι. Does the Commission change its team? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει και αυτή η ομάδα. Ναι. Okay. Good morning. Next is the exchange of views with Willem de Reuter from EMSA. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο De Reuter από την EMSA. Λοιπόν, ξέρω τα μέλη, θα έχω το προνόμιο να επισκεφθώ την ΕΜΤΑ το Δεκέμβριο. Εάν το επιτρέπει ο καιρός, για να πάω να δω την έδρα της εταιρείας στη Λισαβόνα. Έχετε το λόγο για την ενημέρωση όσον αφορά την ΕΜΣΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, να σας πω ότι πετύχαμε το 2010 και ποια είναι η προοπτική για το μέλλον. Είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οργανισμών των μεταφορών και της Επιτροπής αυτής του Κοινοβουλίου πέρσι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έγινε παρόμοια ανταλλαγή απόψεων και αυτό ήταν κάτι χρήσιμο, αλλά και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα να πιστρέψω πολύ πίσω στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα εστιαστώ στα πιο τρέχοντα ζητήματα. Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μόλις τώρα μια πρόταση για την τροποποίηση ε, του βασικού κανονισμού της ΕΜΣΑ, του κανονισμού που δημιούργησε την ΕΜΣΑ υιοθετήθηκε τέλος Οκτωβρίου το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα είναι πρόσφατη η εξέλιξη. Είναι η τέταρτη φορά όπου ο κανονισμός ΕΜΣΑ που υιοθετήθηκε το 2002 ε, τροποποιείται. Κάθε δύο χρόνια λοιπόν φαίνεται να είναι ο ρυθμός που ακολουθείται. Εμπεριέχονται διάφορα στοιχεία στην έκθεση που δεν θέλω να τα αναφέρω όλα. Λοιπόν, η ομάδα, η αρμόδια θα, για τις ρηπάνσεις από πετρέλαιο θα επεκταθεί όχι μόνο να ασχολείται με την ε, ρήπανση ε, που δημιουργείται από τα πλοία και την αυσιπλοεία και βυθιζόμενα δεξαμενόπλια, αλλά πετρελοκυλίδες που επίσης ε, προέρχεται και από ε, υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόριξης κλπ. Λοιπόν, θα πρέπει να διατίθεται ίσως και στις χώρες ε, της πολιτικής γειτονίας τα απορίσματα της ΕΜΣΑ όσον αφορά την ανταπόκριση, την αντίδραση στις ρηπάνσεις να μην βοηθάμε μόνο τις χώρες μέλη, αλλά όλες τις χώρες της Μεσογείου και του ευξήνου πόντου της Μαύρης Θάλασσας. Τρίτο στοιχείο. Η πρόταση υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της υπηρεσίας για την εποπτεία, για θέματα της ναυσιπλοείας, θα πρέπει να είναι κεντρικός ο ρόλος του οργανισμού μας. Και το τελευταίο σημείο προτείνει η τεχνογνωσία της ΕΜΣΑ που έχει αναπτυχθεί για την ασφάλεια, για θέματα ασφαλείας, θα μπορούσε επίσης να διατίθεται και για άλλους τομείς πολιτικής που σχετίζονται, αλλά δεν αφορούν αυστηρά την ε, θαλάσσια, την ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών και μόνο σχετικά θέματα όπως η προώθηση των ε, αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας ε, η εισαγωγή της αρχής e-maritime με ηλεκτρονικό τρόπο δηλαδή για να γίνει πιο, απλούς, ε, πιο απλή η μεταβίβαση ε, διαφόρων εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο η αλλαγή του κλίματος κλπ. Και χαίρομαι να πω ευθύ εξ αρχής ότι έχει, είναι λογική πρώτη. Λοιπόν, Λοιπόν, ένας καλός διάλογος στην προετοιμασία της προσπαθίας ε, περιορίστηκε στην ουσία των διαφόρων ιδεών. Όσον αφορά τον προπολογισμό, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Πάντα ε, ενημέρωνα τους αρμοδίους, υπήρχε πάντα διαφάνεια, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα ε, αντιμετωπίζουμε δύσκολους ε, καιρούς και όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε Υπάρχει κάτι μας Υπάρχει κάτι που όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Σορεύονται όλο και περισσότερα καθήκοντα χωρίς να υπάρχουν προστιθέμενοι πόροι που διατίθενται, χωρίς περισσότερα χρήματα. Μέχρι τώρα μπορούσαμε πάντα να κάνουμε αυτό που έπρεπε, όπως αναμενόταν. Βεβαίως δεν θέλουμε τα αποτελέσματα να υπονομευθούν. αλλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε την ε, σωστή ισορροπία. Κατά τα λοιπά, θα ήθελα να μιλήσω για τα καθήκοντά μας και όχι για τα χρήματα, τη στελέχωση, πόρους γενικά και όλα τα δύσκολα θέματα. Να επιθυμίσουμε ε, τι κάνουμε ακριβώς. Η υπηρεσία έχει πάνω από 20 καθήκοντα, μπορούν να μοδοποιηθούν σε τρεις συστάδες. το πιο, η πιο παλιά συστάδα είναι να δίνουμε βοήθεια, να βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο τομείς για την διενέργεια ελέγχων, να διαπιστώνουμε κατά πόσα κατά πόσο εφαρμόζεται το κεκτημένο για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών και δεύτερον να βοηθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνικώς σε όλα τα ζητήματα που ίσως ανακύψουν. Είμαστε ας πούμε ο σύμβουλος Τη οικογένεια, του σπιτιού. μα καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνουμε τι συμβουλέ όταν χρειάζεται. Ένα καθήκον αυτό, δεύτερο καθήκον. Να δίνουμε βοήθεια στα κράτη-μέλη, αλλά να ενεργούμε σαν πάροχο υπηρεσιών. Να αναπτύσσουμε λοιπόν βάσει δεδομένων για κοινή χρήση από τα κράτη-μέλη. Να αναπτύσσουμε συστήματα για την εποπτεία των θαλασσίων μεταφορών ε, για κοινή χρήση από τα κράτη-μέλη κλπ. κλπ. Και τρίτο καθήκον είναι κάποιες, κάποια άμεσα επιχειρησιακά καθήκοντα ε, τα οποία ανετέθησαν στον οργανισμό κυρίως στον τομέα της ε, ρήπανσης από πετρέλαιο και της αντίδρασης σε περίπτωση ρήπανσης. Θα ήθελα έτσι εν συντομία να επισέλθω σε αυτά τα τρία στοιχεία ξεκινώντας από το τέλος. Δηλαδή πώς αντιδρούμε σε περίπτωση ρήπανσης. Ε, για την ώρα ο οργανισμός μας έχει 15 πλοία που αντιδρούν στη ρήπανση, 15 σκάφη σε μια λυσίδα που είναι στην ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διαμοιρασμένα. Τρία σκάφη στη Βαλτική, δύο στη Βόρεια Θάλασσα, τέσσερα στην δυτική ακτή του Ατλαντικού και πέντε στη Μεσόγειο αντακένα στον εύξηνο πόντο. καράβι. Και την περασμένη εβδομάδα υπογράψαμε και άλλη σύμβαση με έναν φορέα στην Κύπρο αφού έγινε διαγωνισμός και του χρόνου θα μπει σε υπηρεσία και το 16ο σκάφος διότι θα έχουμε νέους πετρελαγωγούς και θα αυξηθεί μεταφορά ε, πετρελαίου από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Όλα τα σκάφη λοιπόν λειτουργούν στα πλαίσια εταιρική συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Η ΕΜΣΑ καθορίζει τι προδιαγραφέ για τα συστήματα ανταπόκριση, αντίδραση σε περίπτωση ρήπανση. Ο κοινοτικό προπολογισμό παρέχει τον εξοπλισμό που θα αγοραστεί, μάλλον τα χρήματα για αγοραστεί ο εξοπλισμό. Τα σκάφη όμως ε, λειτουργούν μέσω ιδιωτικών φορέων. Και καθημερινά κάνουν τη δική τους εμπορική ε, δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή τους αλλά έχουν υπογράψει ε, συμβάσεις αναμονής με την ΕΜΣΑ, άρα αν υπάρξει πρόβλημα σοβαρό με ρήπανση, αμέσως παρατάνε την εμπορική τους δραστηριότητα αυτά τα πλοία και αλλάζουν και γίνονται σκάφη που αντιδρούν στην περίπτωση ρήπανσης και πρέπει πάντα να είναι σε θέση, να είναι σε επιφυλακή, να έτοιμα να αντιδράσουν εντός 24 ώρου αν υπάρξει πρόβλημα και πρέπει να κάνουν ασκήσεις κάθε τρίμηνο και κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε διεθνείς ασκήσεις. Τι κοστίζει τώρα. Χρηματοδοτείται από ένα φακέλο 7 του κοινοτικού προπολογισμού 54 εκατομμύρια 2007 μέχρι 2013 για αυτή την περίοδο 22 εκατομμύρια το χρόνο προβλέπονται από αυτό το ποσό χρηματοδοτούμε και το δίκτυο της καθαρές θάλασσες, Clean Sea Net, που βασίζεται σε δορυφορικό σύστημα για να ελέγχουμε τις θαλάσσιες περιοχές για ρήπανση και όλο το θέμα, όλη η προσπάθεια χρηματοδοτείται από τα 32 εκατομμύρια το χρόνο και για σκεφτείτε, πραγματικά πιάνουν τόπο τα χρήματα ή όχι, εσείς θα κρίνετε. Σύντομα το Κοινοβούλιο θα παραλάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενδιάμεση αναθεώρηση όπως αποκαλείται, διότι 2007 μέχρι 2013 είμαστε στα μέσα του δρόμου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει την έκθεση για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Οι συνάδελφοι μου είπαν ότι σχεδιάζουν να το κάνουν αυτό τον Ιανουάριο και περιμένω την λεπτομερέστερη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Τώρα, αφού μιλάμε για αντίδραση στη ρήπανση, είχαμε το, το γεγονός αυτό, το ατύχημα στον, κόλπο του Μεξικού, που οδήγησε και συζήτηση και εδώ. Κατά πόσο τα πλοία της ΕΜΣΑ θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για να καταπολεμήσουν τη ρήπανση από αυτές τις υπεράκτης εγκαταστάσεις εξόριξης. Ναι, μπορούν. Καταρχήν τα ίδια σκάφη μπορούν να κάνουν και τα δύο καθήκοντα. Όταν η εγκατάσταση υπεράκτια είναι κοντά στις, ε, ε, στους διαδρόμους ναυσιπλοείας, ε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι εκεί τα πλοία ούτως ή άλλως σε αυτή την περιοχή, οπότε δεν κοστίζει πολλά. Αλλά είναι διαφορετικό το θέμα αν αρχίσει να μιλά κανείς για εξόριξη πετρελαίου από πολύ απόμακρες περιοχές, στην Αρκτική ας πούμε, θάλασσα ή αλλού. Καναρίους νήσους, ακτή της Λιβύης ήδη αναφέρθηκαν στον τύπο. Εκεί δεν έχουμε σκάφη που να είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Αν υιοθετηθεί η πρόταση που συζητείτε, θα δούμε. Υποσχέθηκα να μην μιλήσω για, για οικονομικά, για προπολογισμό. Το Δεκέμβριο τα, τα λέμε αυτά. Να μην μιλάμε για αυτά μάλλον το Δεκέμβριο. Το Clean Sea Net ε, το δίκτυο για τις καθαρές θάλασσες. Έχουμε δορυφόρους λοιπόν οι οποίοι μπορούν οι δορυφόροι να ελέγξουν κατά πόσο έχει ρηπανθεί η θάλασσα. Όχι μέσω φωτογραφιών, με ραντάρ. Αν υπάρχει στην επιφάνεια πετρέλαιο, τώρα η αντανάκλαση του ραντάρ αλλάζει και χρησιμοποιεί την αρχή για να δεις αυτή αν υπάρχει ρήπανση ή όχι. Αναπτύχθηκε το σύστημα εκ μέρου όλων των χωρών των παρακτήων της Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Μπορούσαν να αναπτύξουν το δικό του σύστημα ή να ζητήσουν από ένα φορέα να το κάνει ε, για όλους της Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Αυτό αποφασίστηκε και τα κράτη-μέλη το χρησιμοποιούν το σύστημα παραγγέλουν περίπου 2.000 δορυφορικές εικόνες το χρόνο και ε, βάσει τη ζητήσεω κινούμεθα να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία οι παράκτε χώρε και λένε Θέλω να παρακολουθήσω την ε, θαλάσσια περιοχή μου εκεί. Μπορείτε να το κάνετε. Και εμεί κάνουμε τα δέοντα. Μία εικόνα καλύπτει 400 επί 400 χιλιόμετρα. Και τα αποτελέσματα μάλλον βελτιώνονται. Ξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πλοία που περνούν το βράδυ και δημιουργούν ε, κάποια ρήπανση. Στην αρχή είχαμε 1,4 ρήπανση ανά εικόνα. 1,4 ε, επεισόδια ρήπανση ανά εικόνα. Πήγαμε στο 1, 0. Τώρα είμαστε στο 0,86. Ο συντελεστής μειώνεται. Άρα βελτιώνεται η κατάσταση. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Αφού μιλάμε για θαλάσσιο έλεγχο, ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχο, να, πω κάτι και για το Safe CNET. Είναι ένα περιβάλλον κοινών στοιχείων για τον τομέα των θαλασσιών μεταφορών. Κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκαν την ΕΜΣΑ και είδαν ότι σε έγχρωμες οθόνες το σύστημα παρακολουθεί όλη την εμπορική ναυσιπλοεία στις ακτές Ευρωπαϊκής σε όλες τις ακτές. Μπορείτε να, κάνετε, να ζουμάρετε σε μια περιοχή, να κλικάρετε πάνω σε ένα πλοίο και σας δίνει τις λεπτομέρειες για το πλοίο, το σύστημα, όλες τις λεπτομέρειες. Ιδιοκτήτης, σημαία, το λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, εκτιμόμενος χρόνος άφηξης, αν έχει επικίνδυνο φορτίο, ξανακλικάρεις και βλέπεις ποια είναι η φύση του επικίνδυνου φορτίου κλπ. Αν δεν το είδατε, επισκεφτείτε το. Α, θα έρθει ο πρόεδρος να επισκεφτεί. Θα, θα βλέπουμε όλα τα πλοία που πάνε στο Λίβερπουλ, ο πρόεδρος, χαριτολογώντας. Λοιπόν, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από 2.000 διαφορετικές αρχές για τις αλλαγές μεταφορές στην κοινότητα. Συν χίλιες λιμενικές αρχές ακτοφυλακοί, ε, φορείς για το περιβάλλον κλπ. συνδέονται και χρησιμοποιούν τα στοιχεία, δίνουν και πληροφορίες στο δίκτυο και μοιράζονται τις πληροφορίες και αποσύρουν, όχι αποσύρουν μάλλον, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Πολύ πρόσφατα είχαμε νέα εξέλιξη, πολύ ενδιαφέρουσα, που αφορά τα τελωνία. Ανέκυψε το εξής. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε τα ευρωπαϊκά τελωνία για να μπορούν να κάνουν ο διαχωρισμό των πλοίων. Ποια πλοία ασχολούνται με εσωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ενώσης και ποια πλοία έρχονται απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για την ώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Ο τελωνιακός κώδικας λέει ότι οποιοδήποτε πλοίο έρχεται από, εκτός των χωρικών εδάτων των 12 μιλίων προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης και θεωρείται σαν εξωτερικό πλοίο, ακόμα και αν κάνει εμπόριο όμως ενδοκινοτικό. Και είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικά τα τελωνία. Πιστεύουμε με το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο μπορούμε να τους δώσουμε έναν αξιόπιστο τρόπο να μπορούν να κάνουν αυτό το διαχωρισμό, οι τελωνιακοί. Και πριν από δύο μέρες, τρίτη αυτή τη βδομάδα, Έγινε συνεδρίαση ΕΜΣΑ με τι εθνικέ τελωνιακέ αρχέ να συμμετέχουν TG Tax, DG Transport, τη DG Move όπω έχει γίνει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποια ήταν η εντύπωση. Ήταν θετική. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Το 2011 θα ολοκληρωθεί και αν πετύχει μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μείωση διοικητικών διαδικασιών και προώθηση των αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας και ελπίζω και έχω την πεποίθηση ότι θα είναι δυνατόν να γίνει αυτό και θα είναι άριστο παράδειγμα αυτό. Το πώς ένα σύστημα που αναπτύχθηκε απλώς για θέματα ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους χρήσιμους σκοπούς συναφής. Μίλησα πολύ, ίσως. Ναι, το επιβεβαιώνεται. Θα είμαι πολύ σύντομος να πω δύο πράγματα. Έχουμε ένα κέντρο με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα θυμόσαστε σαν μέλη της Επιτροπής των Ιστορικών. Λειτουργεί το σύστημά μας, το ΙΛΑΡΕΙ. Ε, εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη. Αρκετά κράτη-μέλη, ε, μάλλον αρκετά κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισαν να συμμετάσχουν πρώην απικίες, τα Virgin Islands, οι Ολλανδικές Αντίλες κλπ. Το LRTRT είναι το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων στον κόσμο, καλύπτει 25% του παγκοσμίου στόλου. Υπάρχουν 58 τέτοια κέντρα στον κόσμο, επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα, το σύστημα που επιτρέπει την επικοινωνία είναι το International Data Exchange. Το, ανέπτυξαν, ανέπτυξε η Αμερικανική ακτοφυλακή. Μας είπαν οι Αμερικανοί ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν. Για να τα πω πιο σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε να αναλάβει, το ζήτησε ο IMO, ο Διεθνής Αυτιλιακός Οργανισμός και συμφωνήσαμε. Το επεξεργαζόμαστε το θέμα. Το δεύτερο εξάμεινο του 2011 το σύστημα θα μεταφερθεί από την Αμερικανική Ακτοφυλακή, από τους υπολογιστές Αμερικανικής Ακτοφυλακής, στα γραφεία της ΕΜΣΑ στο, στη Λισαβόνα. Και τέλος να πω κάτι για το πιο παλιό καθήκον και το σημαντικότατο, η παροχή βοηθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα μας ε, έκανε οι ομάδες μας έκαναν 83 επισκέψεις ελέγχου το 2010, ολόκληρο φάσμα καλύψαμε, ε, νιογνώμονες, ε, κολέγια, φορείς κατάρτισης για θαλάσσια θέματα και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και σε τρίτες χώρες. Ε, έλεγχος των λιμένων, εγκαταστάσεων των λιμένων. Το σχέδιο είναι να μην αυξήσουμε τον αριθμό των ελέγχων, οι έλεγχοι να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, αλλά να εστιαστούμε περισσότερο ε, σε οριζόντια ανάλυση. Αν έχει γίνει σειρά ελέγχων όσον αφορά τι δυνατότητε υποδοχή των λιμένων, κάποιο πρέπει να κάτσει και να δει τη γενική εικόνα. Ποια μαθήματα μπορεί να αντλήσει από την όλη εικόνα. Τα κράτη-μέλη κάνουν αυτό που πρέπει. Είναι ασαφείς οι κανόνες και πρέπει να αλλάξουν, να ξεκαθαρίσουν τέτοια πράγματα. Συνεργαζόμαστε στενά, αρμονικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση αυτού του χαρακτηριστικού αυτού του στοιχείου. Όπως σας είπα, πέραν των ελέγχων, τακτικά παρέχουμε συμβουλές, είμαστε σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα παραθέσω όλα τα παράδειγματα. Ένα παράδειγμα, εκπομπές είναι θέμα προτεραιότητας. Εκπομπές θείου στη Βαλτική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, που υποχρεωνόμαστε μετά το 2015 να χρησιμοποιούμε πιο καθαρά καύσιμα, πιο ακριβά γίνονται τα καύσιμα, αλλά σχετικά με αυτό το θέμα ανακύπτει και αν υπάρχουν και εναλλακτικές, εναλλακτικά συστήματα. Ε, ειδικά συστήματα για να καθαρίζουν τις εκπομπές αερίου ή καθαριότερο καύσιμο, το υγροποιημένο αέριο πράγματος χάρη. Είναι πολύ και πιο καθαρό και πιο φθηνό. Ε, παρήχθη μια πολύ καλή έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαβιβαστεί. Τέτοια θέματα εξετάζουμε. Αλλαγή κλίματος, διοξείδιο του άνθρακος, δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το μηχανισμό τιμολόγηση, το ETS, όπως και για τις αερομεταφορές ή κάτι διαφορετικό θα χρησιμοποιηθεί. Όποια και αν είναι η απόφαση, οποιο και θα είναι ο μηχανισμός τιμολόγηση, κάποιο θα πρέπει να υπολογίσει πόσο διοξίδιο το άνθρακο παράγεται από κάθε ε, εταιρεία ναυτιλιακή. Και δεν θα με εξέπλητε αν αυτό ο αξέπαινο στόχο στο εγγύς μέλλον καταλήξει πάνω σε κάποιο γραφείο στην ΕΜΣΑ. Ε, αυτά και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω ότι έτσι θα αρχίσει να κυλάει η μπάλα και να ξεκινήσει η διαδικασία αποβολής ερωτήσεων. Ευχαριστώ και ο Ντιρόιτ. Σίγουρα θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Ντερόιτ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Για μας είστε ένας αγαπητός συνάδελφος. Ασχολούμαι με τα θέματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ίσως σήμερα θα είναι η παρουσία σας ευκαιρία να κάνουμε την εισαγωγική συζήτηση ενός θέματος για το οποίο ορίστηκα από την ομάδα μου ως Κιώδης εισηγητής που αφορά τις νέες αλλαγές του κανονισμού και έχω την εντύπωση ότι στη σημερινή σας αναφορά μας δίδει κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα μελετήσουμε περαιτέρω στην ε, παρουσίαση της έκθεσης έγινε από συνάδελφο της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Οι ενδιασμοί που υπάρχουν συνήθως για τέτοιες υπηρεσίες δεν είναι ενδιασμοί που συμμεριζόμαστε για τέτοιες υπηρεσίες. Σωστό είναι αυτό. Διότι η ιστορία, η ιστορία της ΕΜΣΑ εμπλουτίζεται από διάφορα σημαντικά γεγονότα από την αρχή που έγινε ε, με το ατύχημα της Ρίκα, μετά με το Prestige, τα πόσα που διατέθηκαν για τα πλοία τα stand-by και σήμερα ξέρουμε ότι προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγή του σχετικού κανονισμού του 2002. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θα γίνει αυτή η συζήτηση αργότερα. Απλώς θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με θέματα που θέσετε εσεί. Αναφέρατε την καλή δουλειά που έγινε για την ανάπτυξη πλοίων stand-by για, με διάθεση κοινοτικών κολυνδίων 150 εκατομμυρίων. Πρόκειται για πλοία, όχι δικά σας, αλλά τα οποία υπάρχουν εκεί και αιτήσει των κρατών μελών τα βοηθούν σε περίπτωση προβλήματος ρήπανσης. Είπατε ότι έχουμε 15 τέτοιου σκάφη και ετήσι της Κύπρου, όπως είπατε, θα προσθεθεί και το 16ο τέτοιο σκάφος που βρίσκονται σε stand-by, σε κατάσταση επαγρύπνησης δηλαδή. Κατά την άποψή σας λειτουργεί καλά το σύστημα αυτό, αλλά εκφράσατε και ένα παράπονο. Είπατε, σε ποιο μέτρο δεν θα ήταν απαραίτητα και άλλα σκάφη τα οποία θα έπρεπε να πάνε αμέσως σε περιοχές ε, αν συμβεί κάποιο ατύχημα. Φερρυπίν, οι Κανάριες, την οποία έρχομαι εγώ, είναι σε μια ζώνη η οποία δεν προστατεύεται από, αποτελεσματικά από την ύπαρξη σε τέτοια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση των σκαφών που έχουμε τώρα. Κατά πόσον πιστεύετε ε, εσείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να υπάρξει. Επίσης είπατε ότι θέλετε να σας αναθέσουν νέα καθήκοντα. Απ' την άλλη λέτε, τα καθήκοντα θα συνοδευτούν και από ε, οικονομικούς πόρους, γιατί να σας αναθέσουν κάποιος ένα νέο καθήκον χωρίς να σας δώσει το χρήματα για να το φέρει σε πέρας, δεν είναι χρήσιμο. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα αυτό. Επίσης, είπατε ότι αναθέσατε σε μία εξωτερική επιχείρηση την ανάθεση μίας επιθεώρησης. Ξέρω ότι εσείς είστε μία χρήσιμη ε, υπηρεσία και πρέπει όντως είναι προστιθέμενη αξία εάν εσείς αναθέσετε σε κάποιον ε, ε, οργανισμό να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα μπορούσατε κι εσείς αν αυξηθούν οι πόρες σας να αναλάβετε εφόσον είστε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ένα τέτοιο καθήκον. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με το τρίτο πακέτο ρίκα και το λέω εγώ ως ε, ε, Ισπανός στα πλαίσια λοιπόν αυτού του τρίτου πακέτου ίσως θα έπρεπε να δοθούν νέα καθήκοντα στην υπηρεσία σας ώστε να μπορέσετε εσείς να κάνετε περισσότερη δουλειά στα πλαίσια των νέων νομοθετικών πράξεων προβλέπων. Εγώ ήμουν, αν θέλετε, εισηγητής και του οδηγία και του ε, κανονισμού που αφορούσε τους νεογνώμονες. Με την υποστήριξη των ΙΠΑ πρέπει να πω ότι μπήκανε κάποια εμπόδια, αν μπορώ να το πω έτσι, ώστε να μην υπάρχει μηδέα αναγνώριση για τους νεογνώμονες. Πιστεύω ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες νομικής βάσης για να μπορούμε να ενεργούμε όταν έχουμε να κάνουμε με σκάφη τρίτη χωρών. Άρα όντως θα πρέπει να γίνει κάτι όχι μόνο για να μπορούμε να παρέχουμε ε, υποστήριξη και αρρωγή στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις γειτονικές μας χώρες, σε τρίτα κράτη. Θα πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν περισσότερο με αυτό το θέμα. Τελειώνω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε, εάν κατά την άποψή σας, και παρά το γεγονό ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν, οι νέε μεταρρυθμίσει για τους κανονισμούς είναι επαρκής, όχι μόνο για την πρόσθεση νέων καθηκόντων, αλλά πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να τις φέρετε σε πέρας διότι δεν έχετε τους κατάλληλους πόρους. Δηλαδή συγκεκριμένα, Πιστεύετε ότι στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να δοθούν νέοι πόροι στην ΕΜΣΑ για να μπορέσει να αναπτύξει περαιτέρω και τα παρόντα καθήκοντά της και τα μελλοντικά που θα της ανατεθούν. Αυτά μόνο κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάκενστάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ε, του ζητούνται καινούργια πράγματα χωρίς να λαμβάνει νέα κονδύλια για να τα εκπληρώσει. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για τον ε, προπολογισμό, αλλά επίσης πρέπει να πω ότι όσο περισσότερες ε, ε, το ότι σας δίνονται περισσότερες αρμοδιότητες και απαιτήσει είναι, αυτό σημαίνει ότι η ΕΜΣΑ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό ζητούμε και περισσότερα από εσά. Και η ΕΜΣΑ έχει συμβάλει στην ασφάλεια των ε, μεταφορών, στο να βελτιωθεί η ασφάλεια των μεταφορών, να εξελιχθεί. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει και αυτή την ε, θετική αξιολόγηση της Επιτροπής μας να την λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Είπατε επίσης ότι θα υπάρξει ένας ε, νέος αναθεωρημένος κορονισμός για την ε, ΕΜΖΑ, τον, για τον οποίο θα συζητήσουμε ενδελεχώς. Δύο-τρία πράγματα θα ήθελα εγώ να πω, γιατί ούτως ή άλλως ο συνάδελφος είπε πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Πρώτον, το Κοινοβούλιο μετά την ε, καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού με την πετρελαϊκή διαρροή ζήτησε το, να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ. Ερώτημά μου είναι, το χαιρετίζω βεβαίω ότι η ΕΜΣΑ συμμετείχε στις διαδικασίες εκαθάρισης του κόλπου, αλλά δεν θα ήταν πιο σκόπιμο να έχουμε και μια πιο ε, προληπτική προσέγγιση. Δεύτερο ερώτημα. Συγκεκριμένο πάλι. Έχει να κάνει με ένα σημείο σε, αυτό εδώ, σε αυτή εδώ την πρόταση κανονισμού, όπου λέει ότι η ΕΜΣΑ θα υποστηρίζεται ε, περισσότερο από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη ε, σε τέτοιες ε, διεθνείς ε, δραστηριότητες. Εντάξει, αυτό καλό είναι. Ε, δεν δημιουργεί πρόβλημα, το ακούμε να συζητείται ούτως ή άλλως, αλλά θα ήθελα πώς, να μου πείτε πώς ακριβώς θα γίνει συγκεκριμένα αυτό και τι ακριβώς έχει ως στόχο αυτή η κίνηση. Και επίσης ένα πιο διοικητικό θέμα και όχι προς εσάς, ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο. Ε, εκεί στον, ε, στην πρόταση του κανονισμού λέγεται ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο ε, να ρυθμίσουμε τον διπλό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου ως εποπτικό όργανο αλλά και ως εκπρόσωπο αυτών που κάνουν τους ελέγχους. Το πρόβλημα δηλαδή πού ακριβώς είναι. Τέτοιου είδους δομές υπάρχουν χιλιάδες σε όλη την Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λέει η Κομισιόν ότι είναι διπολύπλοκος αυτό ο ρόλο, μήπω μπορεί να μα το εξηγήσει. Ευχαριστώ. Κνούτ, η κυρία Μπιλμπάου. Ε. Καλημέρα σε όλου, Ευχαριστώ τον κύριο Ρόιτερ για τι εξηγήσει που μα έδωσε. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Νομίζω όλοι, όλοι οι υπεύθυνοι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να βελτιώσουμε τις δραστηριότητες μας, να ε, συντονίσουμε τις προσπαθίες μας. Αυτό είναι απόλυτα σαφές, γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε και πιο αποδοτικοί και να είναι και λιγότερες δαπανηρές οι ενέργειάς μας. Αναφέρατε ένα πιλωτικό σχέδιο για να βελτιωθούν οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας. Και ήδη είχατε κάποια συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών για το θέμα αυτό. Εγώ βέβαια συμφωνώ με αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω ότι θα επιτύχει. Αλλά επί αυτού θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, έχετε το ίδιο επίπεδο συντονισμού με την ε, Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, με τη Γενική Διεύθυνση Αλίας, διότι μετά από τις εξηγήσεις που δώσατε πιστεύω ότι στα πλαίσια της αρρωγής σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σημαντικό αυτό που λέω Συνεργάζεστε με την ε, Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, πρώτα απ' όλα για την επιθεώρηση των σκαφών. Διότι εγκρίναμε ε, πρόσφατα ένα κανονισμό για την επιθεώρηση των ε, αλλιευτικών σκαφών. Εσείς είπατε ότι επιθεωρείτε σκάφη, αλλά μας είπατε ότι έχετε ε, τις περίφημες... τους περίφημους χάρτες με τους οποίες με ένα κλικ μπορείτε να δείτε ποια στιγμή ένα αλλιευτικό σκάφος ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος εισέρχεται σε ένα λιμάνι, ε, συντονίζεστε λοιπόν με την Γενική Διεύθυνση Ελίας, τι μάρε. Δεύτερον, αναφέρατε ότι συνεργάζεστε και με την ΙΜΚΟ και αναφέρατε το Κέντρο Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον συντονισμό μεταξύ των 58 κέντρων. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Εσείς συνεργάζεστε με τους υπεύθυνους της επιχείρησης Ατλάντα. Το κέντρο σας μπορεί να προσφέρει μία κάποια βοήθεια σε θέματα πειρατείας. Εγώ δεν είμαι τόσα χρόνια εδώ όπως ο κύριος Γκράντες, αλλά πέρσι στην πρώτη σας παρουσίαση νομίζω ότι αναφέρατε αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας ερωτήσω εάν οι πληροφορίες που συλλέγεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την ΙΜΚΟ μπορεί να βοηθήσει και σε θέματα συντονισμού των προσπάθειων που καταβάλουν την καταπολέμηση της ε, θαλάσσιας πειρατείας στον Ινδικό κενό. Ε, επίσης, σε θέματα ρήπανσης του κόλπου της Βισκάια. Τι συμβαίνει. Είναι υψηλό το ποσοστό ρήπανσης ή είναι σε λογικά επίπεδα. Ευχαριστώ κύριο Στέλλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντερόιτε όχι απλώς κάνετε καλή δουλειά, κάνετε εξαιρετική δουλειά. Οι ομιλία σας ήταν ιδιαίτερως ε, ενδιαφέρουσα και οι προσπάθειες που κάνετε στην ΕΜΣΑ για να μειώσετε τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θείου είναι πραγματικά αξιέπαινες. Κάποια ερωτήματα έχω κι εγώ να θέσω. Προκύπτει από τη δουλειά που κάναμε με, στην Επιτροπή μας με την έκθεση της κυρίας Μάιστες για τον ρόλο της ΕΜΣΑ και το πώς αυτός θα ενισχυθεί. Μιλήσατε για τις ε, πλατφόρμες αντλήσης πετρελαίου offshore που αναφέρονται και στην προτινόμενη θεώρηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς ακριβώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να διαχειριστείτε την αυξημένη ευθύνη και τις συνέπειες που θα έχει ε, η ανάληψη τέτοιων αρμοδιοτήτων και σε χρηματοδότηση και σε προσωπικό κτλ. Δεύτερον, για το θέμα της εποπτείας. Ακούγεται λιγάκι έτσι σαν να είναι μια ιστορία του James Bond με όλες αυτές τις δραστηριότητε, με οθόνες μεγάλες, με δορυφόρους. Αναρωτιέμαι όμως, υπάρχουν, ε, υπάρχει ο εξοπλισμός για να ε, καταγράφονται τα πλοία που που ε, έχουν ε, ε, επιμολυντικό ή επικίνδυνο φορτίο, ειδικά σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές. Και αν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό, γιατί δεν τον είχαμε αξιοποιήσει πιο πριν. Ευχαριστώ. Thank you. Εγώ ευχαριστώ. Πριν να απαντήσω ο κύριος Ντερόιτε, να κάνω και εγώ ένα σχόλιο σχετικά με τις ε, ε, διαδικασίες ε, εκαθάρισης. Θυμάμαι από την αρχή της έναρξης του συστήματος είχαμε κάποια προβλήματα με, παράνομες, με παράνομους καθαρισμούς και θα ήθελα να σχολιάσω το ότι καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό τέτοιων περιπτώσεων. Ε, το καθαρισμό των ε, δεξαμενών ε, πολλοί θεωρούν ότι όταν τον κάνουν στη θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και αποτελεσματική μέθοδος. Ε, βεβαίως εμείς επαγρυπνούμε, ειδικά στην Ευρώπη που έχουμε πολύ ρηχές θάλασσες, πολύ ρηχά εσωτερικά ύδατα και ειδικά στη Βαλτική. Βεβαίως και στις υπόλοιπες θάλασσές μας. Οπότε Εντάξει, είναι μια καλή αυτή αρχή που κάνει η ΕΜΣΑ, μπορούμε, μπορούμε να, να τη χτυπήσουμε στην πλάτη ενθαρρυντικά, αλλά πρέπει να είμαστε, ε, να επαγρυπνούμε και να μην το αφήνουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Ντερόιτε, για να απαντήσετε και μετά η Κομισιόν στο τέλος, εκτός αν θέλετε να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Ντερόιτε, λοιπόν, έχει το λόγο για 10 λεπτά και μετά θα απαντήσει η Κομισιόν. Thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, διότι ήταν σαφέστατες οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω Ετέθησαν ερωτήσεις για την αντίδραση όσον αφορά τη ρήπανση από πετρέλαιο και τις ε, εγκαταστάσεις ε, ε, αντλήσεως πετρελαίου offshore. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο... ποιοι είναι οι παρόντες στόχοι. Ποια είναι τα καθήκοντα που εκτελούμε τώρα. Εντυπωσιάστηκα από τη μνήμη της κυρίας Μπιλμπάου. Ναι, το είπα πράγματι πέρσι ότι θα προσπαθούσαμε φέτος να να καλύψουμε και το βυσκαϊκό κόλπο μέσω ανάθεσης, μέσω συνάψεως σύμβασης με άλλο ένα πλοίο. Και μου λέτε πού είναι το πλοίο. Με θλίψη μου σας λέω ότι ο διαγωνισμός απέτυχε δύο φορές καλέσαμε να υποβληθούν προσφορές. Είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε άλλο ένα πλοίο για την Κύπρο, την περιοχή της Κύπρου και για το Βυσκαϊκό κόλπο. Για την Κύπρο είχαμε καλές προσφορές και Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανάθεσης μας συνέστησε την καλύτερη προσφορά, ποια ήτανε, για το Βυσκαϊκό κόλπο δεν έγιναν προσφορές που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες. Πρόθεσή μας είναι να ξαναδοκιμάσουμε του χρόνου Είναι δύσκολο ο Ατλαντικό κατά κάποιο τρόπο. που προσπαθήσαμε να του ενημερώσουμε, να του ταρακουνήσουμε, να του, πούμε, να πούμε στους υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα προσπαθήσουμε ξανά όμως, του χρόνου. Υπάρχει ανταγωνισμός. Είχαμε το ερώτημα το σχετικό του κ. Γκράμνες, που σωστά το έθεσε, ότι υπήρξε διαμαρτυρία, ισχυρή διατύπωση. Υπάρχει διαμαρτυρία ότι θέλουμε και πλοίο και στις Καναρίους νήσους. Τι κάνουμε γι' αυτό ήταν η ερώτησή σας μάλλον. Για του χρόνου έχουμε εντοπίσει τρεις περιοχές και πρέπει να το συζητήσουμε στην υπηρεσία μας. Με, την, με το Διοικητικό Συμβούλιο το συζητήσαμε το θέμα. Ο Βυσκαϊκός κόλπος είναι στον κατάλογο ο εύξηνος πόντος, έχουμε μόνο ένα πλοίο εκεί και, αυτό, και αυτή η περιοχή είναι στον κατάλογο. Κανάριες νήσι, Δυτική Μεσόγειος και εκεί είναι περιοχές όπου το σύστημα κάπου χωλαίνει πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες και στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεωρήσεως και της εκθέσεως που θα υποβληθεί στην Επιτροπή αυτή ελπίζουμε τον Ιανουάριο θα δείτε το μηχανισμό που εφαρμόζουμε για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, γίνεται ανάλυση κινδύνου και προσπαθούμε να επιδιώκουμε ένα στόχο. Στο μέτρο του δυνατού ακολουθούμε επιστημονική προσέγγιση. Στο τέλος όμως εξαρτώμεθα από τις ε, προτάσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση ε, ρήπανσης από το, από το πετρέλαιο. Τώρα το μέλλον είναι οι μονάδες ε, ε πετρελαίου από το βυθό της θάλασσας, offshore. Κάνουμε κάποιους ενδεικτικούς υπολογισμούς σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για τα συστήματα που έχουμε, για τα συστήματά μας, τι προσαρμογές είναι αναγκαίες και τέλος πόσο θα κοστίσει. Τώρα τι να σας πω. Να σας αναφέρω τους εσωτερικούς ενδεικτικούς υπολογισμούς μας. Απ' την άλλη βέβαια δεν υπάρχουν και μυστικά. Μ' αρέσει να, είμαι, ακολουθώ την αρχή της διαφάνειας. Οι πρώτες ενδείξεις μας δείχνουν ότι υποθέτοντας ότι θα ξεκινήσει στην Αρκτική η ε, προσπάθεια εξόρυξης πετρελαίου και σε άλλες απόμακρες περιοχές όπως είναι οι ακτές της Λιβύης, θα χρειαστούν εν τη αυτή περιπτώσει και άλλα πλοία. Για να το πω απλά, πιστεύουμε ότι το κλασικό έργο στο μέλλον μπορεί να καλυφθεί με το ίδιο ποσό, όπως το παρελθόν, 154 εκατομμύρια για τα 7 χρόνια. Αν μπορεί και αυτό να επεκταθεί, παραταθεί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν επιπλέον έχουμε και το καθήκον των πλατφορμών ε, των υπερακτήων ε, offshore, θέλουμε ένα 10% αύξηση νομίζω. Ίσως να αυτοπυροβολούμε, γιατί ίσως μου πούνε κάποιοι αύριο, αν μου πούνε αύριο μεθαύριο είναι 30% την πάτησα. Τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο είναι ο προβληματισμός. Κάποιο ερώτημα ετέθη για το ζήτημα της πρόληψης όσον αφορά τις πλατφόρμες αντλήσεως πετρελαίου από το βυθό offshore. Ε, είναι κάτι που αναφέρεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι πρόταση, απλώς σαν ένα θέμα προς διερεύνηση και προς προβληματισμό αναφέρεται εκεί. Να πω μερικά λόγια περί αυτού. Αυτές οι εγκαταστάσεις υπεράκτειες δεν είναι το ίδιο όπως τα, τα πλοία του εμπορικού στόλου, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν και ομοιότητες βέβαια. Αυτές οι εγκαταστάσεις, οι offshore, κάνουν γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος. Δεν είναι νησιά, είναι πλωτά, έτσι. Είναι πολύ βαθιά τα νερά, αλλά είναι πλωτές οι δεξάμενες. Είναι ένα είδος πλοίου με ε, ειδικού μηχανισμούς εξοπλισμό για γεώτρηση του βυθού και για άντληση. Οι κανόνες ασφαλείας για αυτές τις εγκαταστάσεις εν μέρη μόνο είναι διεθνείς και καλύπτουν την πτυχή που μοιάζει με πλοίο της εγκατάστασης. Μοιάζουν. Μοιάζει η δουλειά όσον αφορά αυτή την πτυχή. Και ο έλεγχος και η υποπτία γίνεται από τους ίδιους νιογνώμονες. American Bureau of Shipping, Detnos και Veritas κλπ. Και Lloyds βέβαια. Το ξέρουμε γιατί τους ελέγχουμε επί σειρά ετών. Για την αυσιπλοεία. Τώρα αν πάμε στην άλλη πτυχή της γεώτρησης δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε την εμπειρία και εκεί είναι που συμβαίνουν τα τυχήματα όπως είδαμε. Άρα υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ ότι μπορεί το παρόν σύστημα να καλύψει. Μπορεί να καλύψει τώρα και τη γεώτρηση, τη διαδικασία γεώτρησης. Η εταιρεία πετρελαίου ζητά άδεια για να κάνει γεώτρηση και η χώρα που έχει την υφαλοκρηπίδα πρέπει να δώσει την άδεια. Κάθονται λοιπόν οι δύο πλευρές και από κοινού συζητάνε και χορηγείται η άδεια ή δεν χορηγείται. Τι λείπει από τη διαδικασία. Ανεξάρτητος έλεγχος εποπτεί από ένα τρίτο φορέα. Κλασική περίπτωση. Α πούμε για κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, Η διαδικασία είναι συναντώνται δύο ομάδε και ανεξάρτητο τέτοιο φορέα ελέγχει. Και αυτό είναι υποφελέ. Είναι ένα έλεγχο που διεξάγεται. Δεν εξαρτάται από μένα η απόφαση. Δεν μπορώ εγώ να πω κατά πόσο θα απαντηθεί ναι ή ου αυτή η ερώτηση. Οι χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία με τι υφαλοκρηπίδε, το συζητάνε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν η απάντηση τελικά είναι θετική, θα ήταν λογικό να ανατεθεί το καθήκον αυτό στην ΕΜΣΑ. Εγώ δεν βλέπω άλλο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και άλλες γνώσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε και άλλες γνώσεις για το θέμα αυτό. Τώρα, η συνεργασία με την DG Mare. Ο ιδρυτικός κανονισμός λέει ότι εμεί βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό αφορά πάνω από μια γενική διεύθυνση. Η καθήλια αρμόδια όμω είναι η γενική διεύθυνση ε, μεταφορών. Αλλά ήθιστε να συνεργαζόμαστε άμεσα με τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον και τώρα έχει γίνει κλασικό περιβάλλον και κλίμα αυτή η Γενική Διεύθυνση, έχει μοιραστεί στα δύο ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το εξασφαλίσει αυτό, να μπορούμε εμείς να δώσουμε τις γνώσεις μας για να βοηθήσουμε τη διεύθυνση που έχει ανάγκη και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί και κατάλληλη διαδικασία γι' αυτό, για να αποφευχθεί το χάος. Η είναι σε επαφή η τακτική μαζί μας και εμείς με αυτούς. Ρωτήσατε αν τα λιευτικά σκάφη συμμετέχουν στο Safe Net; Όχι ακόμα, σύντομα όμως. Το Safe Net βασίζεται στο AIS, στο αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης. Και τα λιευτικά δεν έχουν πομποδέκτες AIS ακόμα, αλλά από το 2013 και 2014 θα αρχίσουν να έχουν πομποδέκτες. Και τότε θα ενταχθούν πλήρως το LRIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση πειρατεία, ναι. Και χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό. Το κέντρο LRT της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, που εμείς το διαχειριζόμαστε, καθημερινά παρέχει πληροφορίες στη UNAF 4. Και οι στατιωτικοί το χρησιμοποιούν αυτό, χρησιμοποιούν τις πληροφορίε. Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα πλοία με σημαία Ευρωπαϊκή Ενώσεω που μπαίνουν στην καθορισμένη αυτή ζώνη που είναι ευαίσθητη λόγω πειρατεία, αυτομάτω εκεί ενημερώνουμε του στατιωτικού και λέμε να έρχονται αυτά τα πλοία. Και έτσι μπορούν να έρθουν σε επαφή με του ιδιοκτήτε αυτοί και να σχεδιάσουν καλύτερα το πώ χρησιμοποιούν τι φρεγάτε του. Ε, και είμαστε σε συνεχή διάλογο μαζί του. Κύριε Πρόεδρε, τα κάλυψα όλα. Ο κύριος Τέιλορ. Η τελευταία σας ερώτηση. Μου διέφυγε η μισή. Θα είχατε την καλοσύνη σας παρακαλώ να επαναλάβετε. Λοιπόν, αφορά τη χρήση των δεδομένων σας για τις εποπτείας, για τον εντοπισμό επικινδύνων και ρηπαντικών φορτίων. Και αν έχετε τρέξει τέτοια προγράμματα που εποπτεύεται αυτή η δραστηριότητα πλοίων που κουβαλούν επικίνδυνο φορτίο. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Με επιτρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Εμείς παρέχουμε υπηρεσίες μέσω του Safety Net και το χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ένα εργαλείο που ουσιαστικά χρησιμοποιείται για καθημερινό έλεγχο από τις ακτοφυλακές των κρατών μελών. Στην οθόνη λοιπόν μπορούν να δουν οι αρχές αυτές. Κουβαλάει επικίνδυνο εμπόρευμα το πλοίο, ναι ή όχι το σύμβολο που χρησιμοποιείται θα είναι διαφορετικό για αυτό το σκάφος, κλικάρουν πάνω στο επικίνδυνο πλοίο και παίρνουν τι λεπτομέρειε για το φορτίο. Στην ΕΜΣΑ παρακολουθούμε επίση όχι τόσο πολύ για να κάνουν τη δουλειά των ακτοφυλακών, Εμεί παρακολουθούμε να δούμε αν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Εξασφαλίζουμε τη συνέχεια, είναι μια υπηρεσία 24 έως 24, 7 μέρε την εβδομάδα και ελέγχουμε την ποιότητα, αν λειτουργεί το σύστημα κλπ. Αλλά χρησιμοποιείται από τι ακτοφυλακέ. Κατά το παρελθόν συνέβαινε ένα τύχημα. Χρειαζόταν μέχρι και δύο μέρε μέχρι να ξεκαθαριστεί ε, ποια ε, ρηπαντική ουσία διαιρεστεί η θάλασσα λόγω του τυχήματο, αν είναι πετρέλαιο, πετρέλαιο. Βάσει αυτού του συστήματος τώρα γίνεται οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες αμέσως. Όχι μόνο διαθέσιμες για την ΕΜΣΑ, αλλά επιτόπου και για τις αρμόδιες ακτοφυλακές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόσον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ο Ανδρέας Μπόσ είμαι και εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση MOVE. Είμαι ο υπεύθυνος διασύνδεσης με την ΕΜΣΑ. Χαίρομαι που είμαι εδώ και που συναντώ τον κύριο Ντερόιτερ να πω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τον οργανισμό Πράγματι, όπως είπαμε και στην πρότασή μας, θεωρούμε ότι είναι επιτυχής η ΕΜΣΑ και δίνει προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο σχόλιο που αφορά τις συζητήσεις για τις πλατφόρμες offshore, για τις γεωτρήσεις για άντληση πετρελαίου. Να σας παραπέμψω στην ανακοίνωση που δημοσίευσε το Σεπτέμβριο, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η, τη, η Τη Γενική Διευθύνσεως ενέργεια και Αντιπρόεδρο ο κύριος Έτιγκερ δημοσίευσαν αυτό το κείμενο. Το Συμβούλιο έχει καταλήξει συμπεράσματα γι' αυτό και το επεξεργάζεται το θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ανακοίνωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε το τι θα κάνει του επόμενου μήνε για τη βελτίωση τη ασφάλεια αυτών των επιχειρήσεων offshore για την εξόριξη πετρελαίου. Στη DG Move θεωρούμε ότι για την ώρα η ΕΜΣΑ εργάζεται επί της νομικής βάσης για τις μεταφορές. Αν μιλάμε τώρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των offshore, δεν είμαστε πλέον στον τομέα των μεταφορών, χρειάζεται μια συμπροματική νομική βάση και κάτι άλλο. Πριν αποφασίσουμε για έναν οργανισμό όπως η ΕΜΣΑ να κινηθεί στον τομέα τη πρόληψη, θα πρέπει να καθορίσουμε αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σχετικού κανόνε. Πρέπει να πούμε στην ΕΜΣΑ ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιεί για να κινηθεί προς τα χρησιμοποιώντας μέτρα πρόληψης. Τέλος, στο ερώτημα του κύριου Φλέκενστάιν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική για τις επισκέψεις, για τους ελέγχους που πρέπει να δημιουργηθούν από τον οργανισμό. Αν δείτε τώρα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχετε 27 κράτη-μέλη, εκπροσώπου με δικαίωμα ψήφου και 4 εκπροσώπους Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου. Θεωρητικά, θεωρητικά λέω, θα μπορούσε να είναι πολύ περιορισμένη η πολιτική που δεν θα επιτρέπει στον οργανισμό να αναλάβει του ελέγχου όπω εμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμό θα ήθελε να του διενεργήσει. Ε, θεωρητικά αυτή η σύγκρουση ότι υπάρχει σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν άλλα μοντέλα και είδαμε ότι στην ΕΑΣΑ, στην υπηρεσία αερομεταφορών υπάρχει άλλη διαδικασία που θεωρούμε ότι είναι καλύτερη, διότι υπάρχει και επιτροπολογία που έχουν λόγω τα κράτη-μέλη και έτσι έπρεπε να είναι, αλλά η τελική ευθύνη είναι στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί προτείνουμε όσον αφορά αυτό να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη ΕΑΣΑ και να ακολουθηθεί η διαδικασία της επιτροπολογίας και αυτά είναι τα σχόλια που έχω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε καχύποπτοι όταν αναφέρεται η λέξη επιτροπολογία στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ντερόιτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και προσβλέπουμε στην ε, επίσκεψη στις 25 ε, Δεκεμβρίου στην ε, Λισαβόνα. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην υπηρεσία για τους υδροδρόμους ε, και σε άλλους. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα οι κακοί α, ε, της ιστορίας, δεν είμαστε από πάνω για να επικρίνουμε. Το κάνουμε και αυτό, αλλά θέλουμε και να σας διευκολύνουμε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες. Okay, we've covered railways. We've... Ωραία. Καλύψαμε τις θάλασσες, καλύψαμε τα τρένα. Χτες κάναμε τις αεροπορικές μεταφορές, τώρα πάμε στις οδικές μεταφορές, για να δείτε και πόσο πολυσχηδής ομάδα είμαστε. Ο κύριος Πασκαρέλη είναι εδώ, οπότε μάλλον μεταξύ μας θα τα πούμε. Α, είναι και ο κύριος Τέιλορ εδώ. Δύο-τρεις έχουμε μείνει. Ε, να κάνετε την παρουσίασή σας και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Πίτερ, έχει το λόγο. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να σας ε, πω ότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος ε, της Κομισιόν για, το, για τις οδικές ασφάλειες και την ασφάλειά τους, το 2009 περίπου 35.000 ε, άνθρωποι πέθαναν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν και έμειναν με πολλές αναπηρίες. Μπορεί αυτό να συμβεί στο καθένα μας αύριο. Αυτό δεν αναφέρεται στην ε, δημοσιότητα τόσο συχνά. Ε, είναι, εγώ πολλές φορές βέβαια ακούω ράδιο, βλέπω τηλεοράσεις και διαβάζω εφημερίδες και πάντα ε, και κάθε φορά βλέπω έτσι ελάχιστες πληροφορίες γι' αυτό. Βλέπω ε, κυρίως ε, πληροφορίες που αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές. Η πρώτη μου λοιπόν θέση εδώ είναι ότι οι πολίτες μας έχουν, ένα έχουν δικαίωμα σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας των, οδικών, των οδών μας. Γι' αυτό η πολιτική είναι υπεύθυνη, αλλά όχι μόνο η πολιτική. Υπάρχει ε, λοιπόν υποχρέωση και σε σχέση και με τις ε, ε, αεροπορικές μεταφορές ε, δυνατότητα να δράσουμε όλοι. Είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα ευαισθησίας, παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Κατά την ε, λύση των προβλημάτων στις οδικές μεταφορές, η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή η συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της πολιτικής της κοινωνίας των πολιτών, είναι πολύ σημαντική. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός χώρος ασφαλών οδικών μεταφορών ε, και κατευθυντήρες γραμμές ε, για την ασφάλεια του 2000, από το 2011 μέχρι το 2020. Αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε τίποτα αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε η Κομισιόν έγκαιρα πριν εκπνεύσει το τρίτο πρόγραμμα δράσης, που ήδη εδώ και 10 χρόνια ξέραμε ότι θα εξέπνε, να υποβάλει ένα τέταρτο πρόγραμμα. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, ελπίζω να τους ακούσουμε. Κάθε Καθένας που ε, έχει ε, ε, σκοτωθεί ή έχει τραυματιστεί από ένα τέτοιο δυστύχημα ξεπερνάει, πάντα τον, τον αριθμό. Ακόμη και ένας είναι πάρα πολύ. Τα θύματα που διαπιστώνουμε κάθε φορά είναι πάρα πολλά. Προφανώς θα πρέπει να θέσουμε την προστασία των πολιτών μας ως έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Εν τω μεταξύ, και αυτό είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω, είναι ότι πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένου, ε, φιλόδοξους στόχους για τη μείωση αυτών των, των δυστυχημάτων. Πρέπει να έχουμε ενιαίους ορισμού, πρέπει να έχουμε ε, ανταλλαγή, αντικειμενική ανταλλαγή πληροφοριών και υψηλή προστασία δεδομένων. Πρέπει να έχουμε δεδομένους ε, στόχους κοινού μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που τώρα δεν γίνεται ε, υπάρχουν προγράμματα δράση που θα, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Υποστηρίζω την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Κομισιόν, απόλυτα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι οι προτάσεις σε πολλά σημεία δεν πάνε πολύ μακριά, όσο μακριά θα έπρεπε. Ε, νομίζουμε ότι σε κάποια σημεία είναι και, δεν είναι και πολύ συγκεκριμένε και θα πρέπει και μέσω της ε, ε, έκθεσης μου το λέω να γίνουν πιο αντικειμενικοί στόχοι, πιο μετρήσιμοι και πιο χρονικά περιοριστικοί. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει ένα τέταρτο πρόγραμμα δράσης και λευκή βίβλο για τις μεταφορές. Στις, στους 7 στόχους που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν θα έπρεπε να συμπληρωθούν και άλλοι ε, θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει και μια οριζόντια πτυχή και θα ήθελα να πω κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό. Ε, τα μεμονωμένα μέτρα και οι μεμονωμένοι στόχοι είναι σωστοί, είναι σημαντικοί, αλλά χρειάζεται κυρίως ενιαίου ορισμού. Χρειάζονται υψηλά πρότυπα, χρειάζονται δεδομένα, χρειάζονται μέτρα τα οποία να είναι συμπεφωνημένα και να τηρούνται ε, σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί συνάδελφοι ζητούν ε, ε, υπηρεσία ασφάλειας ε, των οδικών μεταφορών. Μια υπηρεσία όπως είχαμε σήμερα το πρωί για τους σιδηροδρόμους, για τις θαλάσσιες μεταφορές. Για, την, για τις οδικές μεταφορές όμως εγώ δεν θα ήθελα να, να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε ένα συντονιστή ίσως ασφάλειας των οδικών μεταφορών, όπως υπάρχει αυτός για, του, για τα δίκτυα TNT ή για τη δημιουργία των, ε, των θαλασσίων περιοχών στο Single ε, European Sky. Μία αρχή δηλαδή η οποία θα μπορεί να συγκερνά τις αρχές των θεσμικών οργανών, τη Κοινωνία των πολιτών, των επιχειρήσεων, ε, των ε, εμπλεκομένων φορέων, να μπορεί να τις συντονίζει και να τις ε, συνδυάζει. Είναι πολλές οι καλές ιδέες που από, και έρχονται από πολλούς φορείς, αλλά δεν τις έχουμε αξιοποιήσει. Για τον στόχο 1, τη δέσμη των μέτρων για τον στόχο 1, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των οδηγών ε, που λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, φυσικά το υποστηρίζω πλήρως. Κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει την ευθύνη που έχει όταν οδηγεί. Και οι οδηγοί των ε, ποδηλάτων και οι πεζοί ακόμη έχουν ευθύνη, από τους μικρούς μέχρι τους ε, ηλικιωμένους. Αυτό πρέπει να το δούμε σφαιρικά. Ακόμη και σε Ακόμη και αυτοί που δεν συμμετέχουν πολύ συχνά, δεν οδηγούν πολύ συχνά, έχουν ευθύνη όταν βρίσκονται στους δρόμους. Και μιλούμε για την ευαισθητοποίηση ε, για τις οδικές μεταφορές. Δεν, ε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν ε, που να πηγαίνει στην να οδηγήσει χωρί να αναλαμβάνει βεβαίω την ευθύνη. Επίσης πρέπει να δούμε το θέμα τη περιποίηση των θυμάτων, των, τραυματιών εφαρμογή ε, των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές. Ε, υπάρχουν αυτά που προτείνει η Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να τα, να τα συμπληρώσουμε. Δεν νομίζω ότι μιλούμε μόνο για την εφαρμογή. Πρέπει να γίνει και μια προσαρμογή, μια ε, εναρμόνιση. Να υπάρχουν συμπεφωνημένοι ομοιογενείς ευρωπαϊκοί κανόνες για, την, για, το, για τα ε, κομμάτια των σιδηροδρόμων που τέμνουν τις οδικές ε, αρτηρίες, ε, για, την, για τις μεταφορές των ε, μεταφορτηγά. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρξει καταστολή όλων των ε, απατών που έχουμε ε, διαπιστώσει στις κατασκευές των οδικών αρτηριών. Θέλω επίσης να εισαχθούν όρια και έλεγχοι ε, όριου ταχύτητας για τον τρίτο τώρα, την τρίτη δέσμη στόχων για τις υποδομές και τις ασφαλείς υποδομές οδικών μεταφορών, ε, οι τεχνολογίες πληροφόρησης, ενημέρωσης, εξύπνα συστήματα μεταφορών θα βοηθήσουν τις ε, υποδομές μας, χωρίς αμφιβολία. Αλλά και με ε, συμβατικά απλά μέτρα, δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, ας πούμε η σήμανση των οδών τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και από τους πεζού και από τους ε, ε, οδηγούς. Ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα υλικά τα οποία, με τα οποία θα επιστρώνονται οι οδικές αρτηρίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με αυτό, επίσης πρέπει να δούμε το θέμα του πάρκινγκ και των σημείων ξεκούρασης στις εθνικές οδούς γιατί ε, και αυτή είναι μια προσέγγιση που αφορά την υγεία, γιατί μόνο κανένας που, έχει, ε, την, ε, που είναι ξεκούραστο και μπορεί να οδηγήσει δεν θα αποτελέσει κίνδυνο στο δρόμο. Επίσης το σύστημα επικούρησης των οδηγών δεν πρέπει να το ξεχάσουμε καλύτερη ε, γενική εποπτεία των φορτηγών, καλύτερες θέσεις για τους οδηγούς αλλά και για τα παιδιά στα αυτοκίνητα. Τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και βεβαίως μετά να, εφόσον έχουμε ε, τέτοια συστήματα τότε που μπορούν να μας εξασφαλίσουν ασφαλή οδήγηση τότε μπορούμε να ξεκουραστούμε να διαβάσουμε την εφημερίδα μας αλλά έτσι όπως οδηγούμε σήμερα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εργαλεία επίσης ε, ε, για την ε, ολοκλήρωση των όρων που υπάρχουν για, τις, για τα οχήματα, λάστιχα, εξοπλισμός που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο. Χτες το κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο ακούσαμε ότι δεν θα, υπάρξει, δεν θα πάρουμε χειμερινά λάστιχα γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που να, τα, που να μας το επιτρέπουν εισαγόμενα προϊόντα όπως ε, αντιλακτικά, ε, λάστιχα, τα οποία δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και αυτά θα πρέπει να τα, να τα ρυθμίσουμε. Ναι, μεν στη, να βελτιώσουμε τα, τις υποδομές μας, ναι, να βελτιώσουμε τα οχήματα, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και τις, ε, και τα τις σωστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε περίπτωση δυστυχήματος. Και αυτό πρέπει να γίνεται και για τα ελαφρά και για τα βαρέα οχήματα. Συστήματα υποβοήθησης όπως το ABS πρέπει να βρίσκονται στον εξοπλισμό, τον, ε, στο στάνταρ εξοπλισμό των ε, οχημάτων και στο στάνταρ εξοπλισμό των ε, φορτηγών. Για την έκτη δεσμίδα μέτρων, αδύναμες ομάδες που συμμετέχουν σε οδικές μεταφορές, βεβαίως υποστηρίζουμε τη ράβωση της Κομισιόν, αλλά πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι ε, ενιαίοι κανόνες για την αντιμετώπιση ε, ατυχημάτων, για τους ε, ποδηλάτες, για τους πεζούς, για τους ανθρώπους σε αναπηρικά καροτσάκια. Επίσης, βελτίωση των δικτών και των δεδομένων. Ποιοτικά δεδομένα, προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε νέε στρατηγικέ. Ίσως να πρέπει να υπάρχει μια βάση δεδομένων για τα ατυχήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργοί θα πρέπει να ε, μπλακούν στην, στο πρόγραμμα δράσης μας. Και κάτι τελευταίο για το σημείο αυτό για τους ε, συγκεκριμένους ε, στόχους που θέλουμε να μειώσουμε το 50% ε, στα τα ατυχήματα κατά 50% μέχρι το 2020. Για τα παιδιά ίσως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να, να, το 50% να γίνει 60%. Προσβλέπω βεβαίως τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας και περιμένω να ακούσω και τις απαντήσεις της Κομισιόν. Στις 7 του Δεκέμβρη θα συναντηθούμε με τον εισηγητή, τον σκιώδη εισηγητή, για να συζητήσουμε όλες αυτές τις ε, πτυχές ε, για να βελτιώσουμε την έκθεσή μου ε, για την, την οποία θα υποβάλω στις 28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ σήμερα και τους συνεργάτες μου και τη γραμματεία και όσους άλλους με βοήθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντέτερ. Η κυρία Σαλάνοβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε μου ζήτησε ο κύριος Τάνια Φάτου, σκιάδες συγγετής, σκιάδες μάλλον, να παρουσιάσω τις δικές της παρατηρήσεις σε σχέση με την έκθεση αυτή. Θα κάνουμε πρώτα απ' όλα μία κριτική της ανακοίνωσης της Επιτροπής, διότι παρά το ότι φαίνεται αρκετά φιλόδοξη, είναι λιγότερο συγκεκριμένη από το προηγούμενο σχέδιο δράσης. Και βεβαίως μείωση κατά 50% των ε, ατυχημάτων ε, για το 2020 είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Αλλά δεν Πιστεύω ότι αυτό είναι το τίμα που πρέπει να πληρώσει κανείς απαραίτητος για την αύξηση κυνηγητικότητας. προβλέπονται προγράμματα αξιολόγησης, επιθεώρησης, τα πλαίσια αυτού του προγράμματος ε, δράσεων, αλλά όλα αυτά είναι γενικότητες και δεν υπάρχει τίτο, τίποτε το συγκεκριμένο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην ε, ε αναθεώρηση αυτού του προγράμματος. Επίσης, δεν βασίζεται καθόλου, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι στα πλαίσια των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών, ε, ποιες θα είναι οι δικές τους δράσεις, ποια είναι η στρατηγική τους, ποιες είναι οι προτάσεις που κάνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές συστάσεις, ήδη πολλές συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του εισηγητού. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ζητήσουμε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες δράσεις που να είναι η βάση των γράφων. Δεύτερον, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής σε συνδυασμό με τα κάθε κράτος μέλος που θα έχει, πρέπει να έχει το καθένα το δικό του σχέδιο δράσης. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και τη διαδικασία αξιολόγησης, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το επόμενο θέμα, καλύτερη συνεργασία σε σχέση ε, με τον ορισμό των τραυμάτων και καλύτερη συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων αστυνομία. Επίσης, αναγραφή της ομάδας αίματος στην άδεια οδήγησης. Επίσης, διασυνοριακή εφαρμογή κάποιων κανόνων και ποιοι, τρί, ποιοι είναι οι αιτίες θανάτου. Η ταχύτητα το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και βεβαίως το ότι κάποιοι δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές, οι πρώτοι συντελεστές των ατυχημάτων. Και βεβαίως πρόληψη και εκπαίδευση μειώνουν τα ποσοστά θανάτων και τραυματισμών. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επιμόρβωση, εκπαίδευση στα κράτη-μέλη, Επίσης, τα έργα υποδομής του οδικού δικτύου είναι σημαντικά και απαραίτητα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την οδική ασφάλεια όχι των κυρίων αρτηριών, αλλά και των ε, δευτερευόντων δρόμων. Ξέρουμε ότι σε κάθε κράτος μέλος επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και προδιαγραφές Άρα η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών δεν μπορεί να γίνει πάντα σωστά, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σωστά στα διάφορα κράτη-μέλη. Ζητούμε λοιπόν να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να έχουμε ως στόχο ασφαλή οδήγηση, ασφαλή οχήματα, ασφαλείς δρόμους. το θέμα της κατανάλωσης ε, υνοπνευματών ποτών είναι πολύ σημαντικό. Η μείωση ε, του ποσοστού υνοπνευματοδών στο αίμα ε, είναι σημαντική, κυρίως για τους επαγγελματίες, οδηγούς, σωστή συμπεριφορά των οδηγών, αμυντική και όχι επιθετική οδήγηση, σωστή εκπαίδευση λοιπόν είναι απαραίτητη. Το πρόβλημα επίσης για τους μεγάλους ειδικίες οδηγούς επίσης τίθεται, διότι η συμπεριφορά τους τα αναγκλαστικά τους είναι διαφορετικά και έχουν μάθει να οδηγούν με άλλες συνθήκες και τα πράγματα αλλάζουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημά τους υπόψη. Ευχαριστώ. Δίτερ. Τέτοιου είδου εκθέσεις είναι η κατάλληλη ευκαιρία να έρθει ο καθένας με το δικό του κατάλογο προτεραιοτήτων. Και έτσι, και έτσι γίνεται σιγά σιγά η οικοδόμηση μια νέα στρατηγική. Έχω εδώ κάνει τι ερωτήσει στο τέλο προ το παρόν, κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την ανακοίνωση τη Επιτροπή θα πω ότι μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Γκρίσμπερκ που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα διότι είχε άλλες σημαντικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Έχοντας αναλύσει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011-2020 σημεριζόμαστε τον κύριο στόχο, μίεση των ατυχημάτων για το 2020 κατά 50%. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι αριθμοί είναι ακόμη πάρα πολύ υψηλοί και πιστεύω ότι επειδή ζητάτε συγκεκριμένα θέματα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιμείνουμε σε τρία θέματα και θα την γνώμη μας είναι πρωταρχική σημασία. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδέα των ελέγχων και των κυρώσεων διασυνοριακά. Θα πρέπει και εδώ να έχουμε εναρμόνιση της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές και να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες. Ίσως, για να δέσω ένα ε, παράδειγμα, θα σας πω τι γίνεται στα σύνορα τα γαλοβασκικά. υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία. Και δεν υπάρχει οι ίδιες κυρώσεις ένθεν και ένθεν των συνόρων. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και στην γειτονική, να την χάνει τις ίδιες προστασίες. Επίσης, το ποσοστό είναι πνευματοδόν ποσών και περιεκτικότητα στο αίμα. Θα πει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθορίσουμε τα ποσοστά. Και, όπως λέει και η ανακλέτες στην ανακοίνωση, θα όπως λέγεται την ανακοίνωση, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες μέρες. Δηλαδή θα μπορούμε κάθε χρόνο με συγκεκριμένο τρόπο να μετρήσουμε το κατά πόσον τα σχέδιά μας μέσω των δράσεών μας ε, υλοποιήθηκαν. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ανατμήματα. Παράδειγμα, και εξηγούμε. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα οδικής ασφαλείας οι νεαροί που καταναλώνουν πολύ περισσότερο αλκοόλ με τους επαγγελματίες οδηγούς και με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Δεν μπορούμε με γενικούρες να βρίσκουμε λύσεις. Επίσης, τα βαρέα οχήματα είναι το 3% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι υπεύθυνα για το 14% των ατυχημάτων και σε κάθε κράτος μέλος προκαλούν 4.000 θανατηφόρα, ε, ε, θανάτους, ε, θανατηφόρα ατυχήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η δική τους ευθύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό συγκεκριμένα. Να δούμε επίσης πώς θα μπορούσαμε τέτοιου είδους ε, οχήματα να τα βελτιώσουμε, έτσι θα δημιουργήσουμε και νέες θέσεις απασχόλησης στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Δηλαδή, εφόσον αυτά τα μεγάλα φορτηγά δημιουργούν τέτοια οχήματα, να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε φερρυπίν, μειώνοντας τα τις μαύρες επιφάνειες όπως λέμε, δηλαδή το κομμάτι που δεν μπορεί να μπει δει από τον ε, ε, καθρέφτη του οδηγός ώστε να μειώνονται τα ατυχήματα. Τα θέματα λοιπόν της οδικής ασφάλειας είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να χειριστούμε από την αρχή, από την κατάρτιση, από την ε, παιδεία των παιδιών, ώστε σιγά σιγά δεν αρκούν μόνο να έχουμε ε, διαφημίσεις, να μαθαίνουμε σιγά σιγά στα παιδιά ώστε να αποκτήσουν την οτροπία ότι πρέπει να είναι ε, πιο προσεκτικά. Στο το θέμα των ελέγχων, η έλεγχοι που γίνεται στους αυτοκινητοδρόμους, ε, λέγονται κάποια αλλά όλο και περισσότερο αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν με τρομερές ταχύτητες έχουμε γύρω μας και έτσι κάποια στιγμή χάνουμε και την αίσθηση, ε, κάνοντας συγκρίσεις, χάνουμε την αίσθηση της ταχύτητας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μην συμπεριλάβω εγώ το δικό μου κατάλογο επιθυμιών. Γενικά θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των τραυματισμών και των θανάτων στους δρόμους και είναι μια κατάρα σύγχρονη και έχει κοινωνικές συνέπειες. Το ανέφεραν και άλλοι ε, μέλη. Έχουμε συνέπειες αυτά και για τις ε, υπηρεσίες περίθαλψης. Ε, κοστίζει λοιπόν και οι θάνατοι κοστίζουν. Γενικό κόστος λοιπόν λόγω των ατυχημάτων. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας να συμπεριληφθούν ε, και διάφορες ε, ευάλωτες ομάδες. Δεν ξέρω αν μπορούμε τελικά να τα αποκριθούμε στις ε, προσδοκίες βασιζόμενοι στα FEE e αυτοκίνητα. Αναφέρθηκαν και άλλοι στις υποδομές, ανησυχίες που έχουν. Μπορούμε να βρούμε ποια είναι τα κενά του εγγράφου Υπάρχει αναφορά της συνθήκης της Αβώνας συγκεκριμένη, όπου έχουμε το άρθρο 90, το οποίο θέτει ευθύνε όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Στα χέρια μας θέτει αυτό το, το καθήκον. Χρειάζεται και καλύτερος έλεγχος των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους 130 χιλιόμετρα την ώρα, σε αστικές περιοχές 30 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των ε, εξαιρέσεων που θεσπίζει η τοπική αυτοδίκηση. Το ενόπνευμα, βασικό αίτιο ατυχημάτων, ε, πρέπει να υπάρξει ένα κοινό όριο που θα επιβάλλεται παντού, σε όλη την Ευρώπη. Κανένα ναρκωτικό, κανένα φάρμα, κανένα ναρκωτικό μάλλον δεν πρέπει να καταναλώνεται από τους ε, οδηγούς και όλα αυτά με τα όρια ταχύτητας δεν είναι θέμα εάν πρέπει ή όχι και επίσης ε, και ε, όσον αφορά τη χρήση νοπνεύματος Πολύ λίγοι νέοι ε, πίνουν και οδηγούν, αλλά αυτό δεν είναι μαύρη παρηγοριά ένας έχει πατήσει αυτοκίνητο. Πρέπει να καλύπτουμε τους πάντες με την νομοθεσία μας. Παρόλο που όσον αφορά το όριο για την κατανάλωση νοπνεύματος θα καλύψει μόνο ένα ποσοστό. Και επίσης υπάρχουν και κακές περιοχές, επικίνδυνα σημεία στους δρόμους Ευρωπαϊκής Ενώσης. Πρέπει να τα βελτιώσουμε αυτά τα σημεία και αν αυτό είναι ανέφικτο, πέραν από την επιδίωξη βελτίωσης πρέπει να ενημερώνουμε τους χρήστες των οδών. Χρειάζονται εκστρατείες για ενημέρωση, για βελτίωση ασφάλειας για ομάδες χρηστών, για ποδηλάτες, για πεζούς, κυρίως για ευάλωτους, ε, ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι και οι χρήστες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Ε, υπάρχει ανησυχητική τάση και εκεί. Και νέοι που οδηγούν τα Σαββατοκύριακα και μόνο. Και αυτοί προξενούν ε, δυσανάλογα πολλά ατυχήματα. Τέλος, ας μην λησμονούμε την ανάγκη να προωθήσουμε αλλαγή νοοτροπίας και μοντέλων. Να μην χρησιμοποιούνται τρόποι μεταφοράς που βλάπτουν το κοινοβούλιο, αλλά πιο βιώσιμες μέθοδοι μεταφορών, τρένα, λεωφορεία, ποδήλατα, βάδισμα. Σαν σκιώδης των Πρασίνων σε αυτό το θέμα θα ήθελα αυτή, αυτά τα θέματα, αυτή η θεματική να προωθηθεί. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντίτερ Κοχ για την ε, πολύ καλή έκθεση του περιληπτική. Είναι πολύ περίπλοκο και το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών και νομίζω ότι προχωράμε μεγαλύτερο θάρρος από ό,τι η Κομισιόν στο, όταν, θα υποβληθεί το εγγραφό του, η εκθεσή του θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες για να το διορθώσουμε εδώ και εκεί, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το α, συζητήσουμε γενικώ, γιατί η ασφάλεια των μεταφορών αφορά όλους μας και οι φιοντοφορές έχουν γίνει και διασυνοριακό θέμα. Οπότε και εμείς καλό είναι που ασχολούμαστε με ένα τέτοιο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα για τα μεμονωμένα στοιχεία, ο Ντίτα το είπε ήδη, πρέπει να δούμε την ευθύνη του κάθενό. Βεβαίω θα χρειαστεί έτσι και περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό. Νομίζω ότι παλαιότερα υπήρχε στην ε, η γερμανική τηλεόραση μια εκπομπή ειδική για την, ε, για την ασφάλεια των ε, οδηγών και είναι, έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει στην ευθύνη και στην ε, ενσυνείδητη οδήγηση των γερμανών οδηγών. Δυστυχώ αυτή η εκπομπή κόπηκε πια και δεν τη βλέπουμε. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την αύξηση των μεταφορών. Ε, η Ευρώπη τόσο άλλως είναι χώρα διαμετακόμισης για πολλά αγαθά που περνούν από εμά και μετακινούνται. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την εξίσωση των ε, κανόνων. Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις ε, οδήγησης για να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει τους κανόνες που ισχύουν στις υπόλοιπες ε, χώρες, <coughs> τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Μπορώ να σας πω πολλά περί, παραδείγματα από το Βερολίνο. Κάποτε δεν είχαμε τραμ, τώρα έχουμε. Και ο κόσμος ε, κυκλοφορούσε ε, με το ελεύθερα κάποια στιγμή που, ξέ, που δημιουργήθηκε το τραμ ε, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά δυστυχήματα γιατί ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει να περπατάει στο δρόμο και εκεί που παλιά περπάταγε εκείνη, μετά υπήρχε το τραμ οπότε υπήρξε μεγάλη, μεγάλη, υπήρχαν πάρα πολλά δυστυχήματα. Το πώς συμπεριφέρεται κανείς στην ε, κυκλοφορία βεβαίως είναι δική του ευθύνη. Και οι αριθμοί στην ε, Γερμανία δείχνουν ότι στον, ε, στον αυτοκινητόδρομο που δεν υπάρχει όριο ταχύτητα ε, δεν είναι κατά ανάγκη πιο υψηλά τα δυστυχήματα από ότι είναι σε οποιοδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε άλλη ειδική αρτηρία. Ευχαριστώ κύριε Ζέλερ. Να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα πριν περάσουμε στο όριο ταχύτητας ή στην έλλειψη ταχύτητα η στην ελλειψη οριου ταχύτητα στη γερμανια ειναι εξαιρετικη η εισαγωγή που κάνατε κύριε, κύριε Κόχ. Φαντάζομαι ότι και με τους ε, σκιώδεις θα γίνει μια πολύ καλή πρόταση. Ε, νομίζω ότι ήσασταν τότε μέλος του Κοινοβουλίου. Είναι λίγο σαν να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Όταν είχαμε την έκθεση της κυρίας ε, Πίτερσεν πριν από κάποια χρόνια. Και ίσως καλό θα ήταν να τη δείτε, να δείτε τι είχε γράψει τότε, πριν από 8-10 χρόνια είναι σαν, σαν να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο από την αρχή. Από που λέγαμε, σε σχέση με αυτά που λέγαμε τότε. Χαμηλό αλκοόλ, όρια ε, ταχύτητας, όλες οι επιθυμίες που έχει κανείς, τα είχαμε πει και τότε. Οπότε, ίσως, στην, ε, για την έκθεσή σας, θα άξιζε τον κόπο να ρίξετε μια ματιά και σε αυτή την ε, έκθεση. Δύο παρατηρήσει να κάνω εγώ. Κάποιο μίλησε για τα έξυπνα αυτοκίνητα. Χρειαζόμαστε έξυπνη, έξυπνα αυτοκίνητα γιατί δεν έχουμε έξυπνου οδηγού. Αυτό είναι το κακό. Οποιοδήποτε προσπαθήσει να πάει σπίτι του, προσπάθησε να πάει σπίτι του χτες, ε, θα ήταν, ήταν απόλυτο παράδειγμα ε, μη έξυπνο οδηγού προσπαθώντα να οδηγήσει μέσα στο, ε, μέσα στο χιόνι με τα λάθο λάστιχα, με λάθο νοοτροπία. το ίδιο κάνουμε ε, το ίδιο, ε, με τον ίδιο τρόπο οδηγούμε την 1η του Δεκέμβρη και με τον ίδιο τρόπο οδηγούμε την 1η του Ιούνιου, ανεξαρτήτω καιρικών συνθήκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Να πω και κάτι που το είπαν και οι υπόλοιποι. Εφαρμογή. Μπορούμε να έχουμε του καλύτερου νόμου του κόσμου. Αν δεν εφαρμόζονται, είναι άχρηστοι. Το είπατε κι εσείς βέβαια στην εισαγωγή σας. Ένα ακόμη θέμα που είναι στις δικές μου επιθυμίες. Ε, τι γίνεται με, τα, με, τις, δια, με τις διαβάσεις, ανισόπεδες διαβάσεις. Τι κάνουμε όταν κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να περάσει την ε, σιδηροδρομική διάβαση από την ανισόπεδη διάβαση. Εγώ έχω δει πολλούς ανθρώπου να το κάνουν κάθε μέρα ακόμη και με παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Να, έχουμε, να υπάρχουν ε, που κατεβαίνουν στις ε, γραμμέ για να μην μπορεί να περάσει κανείς. Ίσως αυτό είναι μια λύση. Ίσως μια λύση να είναι ένα χρηματικό ε, πρόστιμο. Και κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να επενέσω τις, γερμανικές, τις γερμανικές αρχές είναι οι ρυθμίσεις που υπάρχουν ε, στους, ε, στα τιμόνια των, ε, των βαρέων οχημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι αν ένα φορτηγό έχει βάλει νέα ελάστιχα και πάθει κάποιο πρόβλημα στο δρόμο και πάει με τις άντες για 400 μέτρα, αυτό που γίνεται είναι ότι βγαίνει ε, το λάστιχο, μπαίνει ένα νέο λάστιχο και δεν υπάρχει καμία εποπτεία, κανένα έλεγχο για το αν έχει, έχει πάθει κάποια ζημιά η Ζάντα ή οτιδήποτε. Μόνο οι Γερμανοί έχουν σύστημα εποπτείας και το ελέγχουν αυτό. Ας δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα του πώς αλλάζουμε τα λάστιχα, τι γίνεται με τις ζάντες σε περίπτωση ε, ατυχημάτων και θα πρέπει να σταματήσουμε να, ε, ε, αυτό, το, αυτή τη συνήθεια που υπάρχει, να βάζουμε λάστιχα σε χαλασμένες, καινούργια λάστιχα σε χαλασμένες ζάντες. Γιατί νομίζω ότι το είπε και η κυρία Μπιλμπάου. Πολλά από τα ατυχήματα γίνονται από βαρέα οχήματα. Οι περισσότεροι είναι οδηγοί σε καλέ ε, εταιρείε βέβαια, αλλά αν πάει κάτι στραβά, τότε σίγουρα κάποιο άνθρωπο θα την πληρώσει. Η Κομισιόν τώρα. Ο κύριο Πασκαρέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοχ και όλους τους συναδέλφους σας που συμμετείχαν στη συζήτηση. Δεν θα Περιγράψανε εκείνες της Επιτροπής. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά την παρουσίαση με εύλατο τρόπο ο κύριος Κόχ. θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Συζητάτε σήμερα αυτό το θέμα και συγχρόνως το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών προσπαθεί να συμφωνήσει για την πρόταση της για την εφαρμογή των ε, προβλημάτων που δημιουργούνται στα ανισόπεδες διαβάσεις περιλαμβάνονται στις ε, γενικές γραμμές πλαίσης Κομισιόν. Από μεριά μας έχουμε τεχνικούς εμπειρογνώμονες για στατιστικές και συλλογή δεδομένων που αφορούν την οδική ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παράγουμε μόνο γενικόλογα έγγραφα, αλλά η δράση μας συνεχίζεται καθημερινά. Βεβαίως έχουμε τα όρια μας και τους περιορισμούς μας στο τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως σε επίπεδο Επιτροπής για την Αδική Ασφάλεια. Έχουμε όμως και ευκαιρίες. Οι περιορισμοί μας ποιοι είναι. Πρώτα απ' όλα, ήδη πολλά έχουν γίνει σε θέματα νομοθεσίας και δράσης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν σε αυτών. Σε επίπεδο διεθνέ στο επίπεδο τη οικονομική και κοινωνική επιτροπή του ΟΗΕ, στα πλαίσια της Σύμβασης της Βιέννη για τον κωδικό, κωδικούς ασφαλείας του δικού Ήδη λοιπόν έχουν γίνει πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τώρα την νομοθεσία, αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε νέα νομοθεσία. Δεύτερος περιορισμός. Η περίφημη επικουρικότητα περισσότερο από σε άλλους τομείς, στον τομέα των μεταφορών, η επικουρικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο για την ε, ευθύνη που φέρουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε κράτος, αλλά στην ευθύνη του κάθε κράτους και σε εθνικό και παραπέρα, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και οι δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή η ευθύνη του καθενός για τους ανασφαλείς δρόμους, για το τίμημα που πληρώνουμε με τις ζωές μας και θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει συλλογικά και όχι μόνο η Κομισιόν να κάνουμε κάτι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το τόσο ε, φιλόδοξο στόχο μας. 2020 μείωση των θετηφόρων ατυχημάτων 50%. Μπορεί να μην φτάσουμε το 50%, το 40%, αλλά σίγουρα 100.000 ζωές θα σωθούν, αν όχι περισσότερες. Η επικουρικότητα επίσης, αν πάρει τα πράγματα από τη διαφορετική σκοπιά, μία ευκαιρία. Διότι είναι πάλι μοιρασμένη ευθύνη για όλου. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένα πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνο για την οδική ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα, επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάποια από τα ειδικά σχόλια που έκαναν οι συναδελφοί σας. Δεν θα απαντήσω σε κάθε θέμα που αφορά ε, αυτά που ισχυριστήσετε για την shopping list, τις επιθυμίες του καθενός. Το θέμα των ορισμών και των προδιορφών. Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά ήδη πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει πολλά. Μόλις τώρα δημοσιεύθηκε ένα ειδικό εγχειρίδιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές πληροφορίες μετά τις έρευνες που κάνατε. Έχουμε μία βάση δεδομένων που λέγεται CARE, η οποία δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε μετά από μία απόφαση των ε, υπουργών ε, από τη δεκαετία του 60-70, που είναι ένας θησαυρός δεδομένων για τα οδικά ατυχήματα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα, και αυτό είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχουμε στις γενικές γραμμές πολιτικής που ακολουθήσουμε, είναι ένα τρόπος αμερόληπτης ερεύνησης των οδικών ατυχημάτων όπως κάνουμε και για την, ε, οδική, για την ε, σιδηροδρόμους και για την ε, ναυσιπλοεία. Πολλοί λοιπόν ζητούν και εσείς και ενδιαφερόμενοι άλλοι φορείς τη δημιουργία ενδεχομένω μιας υπηρεσίας ασφαλείας όπως έχουν οι σιδηρόδρομοι και τα πλοία. Πρέπει να σας πω ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι τεχνικές υπηρεσίες που υποβοηθούν την Κομισιό για, ε, για να λάβει κάποιες αποφάσεις και αναφέρουμε σιδηροδρόμους στην αεροναυτιλία και στην αυσιπλοεία, αλλά για, τις, για ε, την οδική ασφάλεια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ποια είναι η διαφοροποίηση της οδικής ασφάλειας από την ασφάλεια άλλων τρόπων μεταφορών. Πόσο σημαντικό είναι το ανθρώπινο στοιχείο, η εκπαίδευση, η συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα. Πολύ περισσότερο εδώ επισέρχεται το στοιχείο άνθρωπος από ότι στα άλλα είδη μεταφορών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το προβλέπουμε στις δικές μας γενικές πλεύσεις και βεβαίως αφού έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία θα πρέπει οτιδήποτε γίνει να γίνει και να ισχύσει και σε εθνικό επίπεδο. Διότι τώρα, όπως είπε και ο κύριος Τέιλορ, με την συνθήκη της Λισαβόνας αρχίσουμε να έχουμε μια κάποια ευθύνη κοινοτική, υπάρχει δικαστική αστυνομική συνεργασία, και βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο την οδική ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια όλων των μεταφορών των οδικών, δηλαδή όχι μόνο τα, των οδιωτικών οχημάτων. Επίπεδο πνεύματος, στο αίμα, η τροχή, η κατάλληλη τροχή, η ταχύτητα. Αναθερούμε και την σχετική νομοθεσία τώρα για την καταλληλότητα των τροχών. Πρόκειται για μία οδηγία η οποία αφορά την καταλληλότητα και την ασφάλεια των τροχών των αυτοκινήτων και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ώστε επιτόπου να υπάρχει με καλύτερη ευθύνη και συνειδητοποίηση των κινδύνων. Και βεβαίως ε, υπάρχει το θέμα τη κανόνα που ισχύουν για την οδική ασφάλεια στο χώρο στον οποίο ε, πληρώνεται τις, ε, τα τέλη κυκλοφορίας αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος έλεγχος αλλού ώστε να μπορούν να γίνονται ε, τέτοιου είδους έλεγχοι και εκτός των χωρών στις οποίες έχουν ε, ε, γίνει, γίνεται η θέση κυκλοφορία του αυτοκινήτου και να γίνεται αυτός ο έλεγχος καταλληλότητας των οχημάτων. Αλλά αυτό απαιτεί και περισσότερη ε, συνεργασία. Ακούστε, η οδική ασφάλεια τώρα δεν είναι κάτι το μεμονωμένο στα πλαίσια της πολιτικής μας, έχει σχέση και με όλα τα θέματα που αφορούν τις μετακινήσεις, τις μετακινήσεις για όλους γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σφαιρική η προσέγγιση μας. Μία απάντηση στην κυρία Μπιλμπάο. με τις ε, παρατηρήσεις τις οποίες συμφωνούμε απολύτως. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι ε, και να μην έχουμε μία σφαιρική λύση ε, για κάποια θέματα. Θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Και μίλησε και το επίπεδο υνοπνευματοδών, ε, ποσοστού πνεύματος στο αίμα. Έχουμε εδώ κάποια θέματα από αυτά που είπατε, τα οποία συμπεριλάβαμε στον εγχειρίδιο αυτό καλών πρακτικών. Και είπατε ότι θα πρέπει να ορίσουμε διαφορετικά επίπεδα περιεκτικότητα συνοπνεύματος στο αίμα ανάλογα την κατηγορία του οδηγού. Νέου, επαγγελματία κτλ. Είπατε η κυρία Μπελμπά σωστά ότι τα φορτηγά είναι υπεύθυνα για 14% των ατυχημάτων. Πρέπει να κάπως να το διορθώσω το θέμα. Εμπλέκονται κατά 15% τα φορτηγά σε τέτοιου είδου ατυχήματα. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι σε τόσο ποσοστό και υπεύθυνα για το ατύχημα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν εμπλέκεται ένα φορτηγό σε ατύχημα, τα πράγματα είναι διαφορετικά από το να έχει γίνει ατύχημα μεταξύ δύο μικρών smart. smart. Το... Για νησόπαιδες διαβάσεις. Το θέμα της ασφάλειας ε, για τη... 700, 600. Των διαβάσεων είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και εμάς υπήρχε και έτος ειδικό το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να πω ότι η διάβαση των ανισοπαίδων, το πέρασμα των ανισοπαίδων διαβάσεων είναι στατιστικά ο μεγάλος υπεύθυνο ε, και για τα ατυχήματα που καταγράφουν οι σιδηρόδρομοι. Και βεβαίως, όπως είπατε, η εκπαίδευση, η παιδεία, η κατάρτιση για να εφαρμοστούν οι πολιτικές και η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά αποτελούν σχέδιο δραστηριοτήτων, ένα action plan που θα αναλάβουμε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει και έναν από τους στόχους προς Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δίτε μπορεί να το ελέγξεις αυτό. Είναι ε, απίστευτα τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε αυτές τις διασταυρώσεις στη διαλευση των τρένων, στις ισόπεδες διαβάσεις. Ε, να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους και τις προτάσεις τους. Δεν είναι κατάλογος ε, ε, του σούπερ μάρκετ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι δώρο Χριστουγέννων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι. Ε, χαίρομαι που συμφωνούν και οι άλλοι μαζί μου ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Βεβαίω να δούμε και τη συζήτηση για την επικουρικότητα. Ε, πρέπει λοιπόν κάποιο να πάρει το θάρρο και να πει ποιο είναι ο υπεύθυνο τελικά. Όλοι κοιτιόμαστε και τελικά κανένα δεν, δεν αισθάνεται υπεύθυνο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναλάβει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πολύ σωστό αυτό που είπατε στο τέλος. Ε, ευχαριστώ, Ντίτερ. Το σχέδιο έκθεσης θα αποβληθεί στην Επιτροπή το Φεβρουάριο, θα ψηφίσουμε τον Μάιο και στην Ολομέλεια του Ιουνίου μετά για να έχετε μια γενική εικόνα. Ξέρω ότι υπάρχει συνάντηση σκιωδών εισηγητών με τον εισηγητή την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Έξοχη συζήτηση. Στα διάφορα να σας ανακοινώσω ότι έχουμε δύο μέλη, ο Βάλερη Χίλτης Βίφτη, επίσης κύριε Βίφτη, αποχωρούν. Έκανα πρόβες επί 20 λεπτά και ακόμα ε, πάλι, πάλι δεν τα κατάφερα. Ζητώ συγγνώμη αν δεν ανέφερα το, στο όνομά σας. Ε, πάνε σε καινούργια δουλειά. Ο Γιώργο Ντίτχαρτ καταφθάνει σε καινούριο μέλος. Τον έστειλε η Ντόρις Πακ από την Ολέα Πολιτισμό και Αθλητισμό. Καλώ ήρθε. Βάλερη και Ζιβίλ, ό,τι καλύτερο στα νέα σα καθήκοντα. Να σας πω συνάδελφοι ότι η επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις 3. Άρα πρέπει να σας ευχηθώ σε όλους. Δεν πρέπει, θέλω να σας ευχηθώ. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο τον νέο χρόνο και αυτό ισχύει μόνο για τους βουλευτές και για τους βοηθούς όλους τους έρχοντες στην Επιτροπή και τέλος, εξίσου σημαντικό αυτό, και τους διερμηνείς απευθύνω τις ευχές, χωρίς τους οποίους εγώ θα είχα κάποια προβλήματα σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας.